On va commencer. Mesdames et messieurs. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Σιγά σιγά κυρίες και κύριοι, ξεκινήσουμε. Ah Alors, euh, d'abord. Λοιπόν, καταρχήν, μια διευκρίνηση για τους πολυάριθμους βουλευτές που ήταν εδώ το πρωί. Υπήρξε μια παρεξήγηση το πρωί για ένα επιπλέον σημείο που προσθέσαμε στην ημερήσια διάταξη, δηλαδή την ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες για την έκθεση του κυρίου Σβένσον για, για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Η γραμματεία μου ζήτησε να διευκρινίσω τα εξή. Αυτό το επιπλέον σημείο αρχικά το ζήτησαν οι πράσινοι, αλλά πριν από πολύ καιρό. Μου έγινε κάποια παράληψη στη γραμματεία και δεν προστέθηκε στην ημερήσια διάταξη. Προσπάθησε η γραμματεία να διορθώσει το λάθο και το, προ... πρόσθεσε στη σημερινή ημερήσια διάταξη, αλλά αυτό δυστυχώ ανακοινώθηκε μόλι σήμερα το πρωί στην αρχή τη συνεδρίας τη Επιτροπής μα. Αυτό δημιούργησε κάποιε δυσκολίε σε ορισμένου βουλευτέ που δεν κατάφεραν να είναι παρόντε. Άρα η ευθύνη για την παρανόηση δεν είναι ευθύνη καμιά πολιτική ομάδα, γιατί εγώ σήμερα το πρωί δεν καταλάβαινα γιατί πράσινοι ένα σημείο και δεν ήταν παρόντες. Τώρα ξέρουμε. Επίσης, μια μικρή τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη, η ανταλλαγή απόψεων για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματο Εθελοντών για την επιστηστική βοήθεια θα είναι μετά το σημείο του κυρίου Γκέρεν για το ΣΑΧΕΛ, γιατί θα πρέπει να φύγει ο κύριο Γκέρεν στη συνέχεια. Αλλά δεν είναι καν εδώ ο κύριο Γκέρεν. Θα έρθει, εν πάση Έχετε όλη την κάρτα σας για την ψηφοφορία. Εγώ παραλίγο να την ξεχάσω τη δική μου. Αλλά δεν ήθελα να γίνω ρεζίλη, να μην έχω την κάρτα μου. Ας ελέγξουμε λοιπόν. Δεν έχω την κάρτα μου, Πρόεδρε. Θα μας κεράσετε σαμπάνια στο τέλος της συνεδρίασης. Κάβα, καταλανική σαμπάνια θα σας κεράσουμε. Λοιπόν, για τον κύριο Κερέρα θα κάνουμε μια εξαίρεση και θα δεχθούμε χωρί κάρτα την ψηφοφορία του, αλλά με τη σαμπάνια στο τέλο τη συνεδρίαση. Α κάνουμε τη δοκιμαστική ψηφοφορία. Μας λείπει κάποιος? Μήπως κάποιος ξέχασε να ψηφίσει? Μας λείπει ένας. πέρα της ψηφοφορίες. Ωραία. Ας αρχίσουμε. με την έκθεση Μπέρμαν. Μισό λεπτό. Ήξερα ότι κάτι μου διαφεύγει. Ωραία, τώρα έχω και τα ακουστικά μου. Προτείνω να ψηφίσουμε μαζί για την έκθεση του κυρίου Μπέρμαν on block. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Le vote est clos. Πέραση της Homophone Ομόφωνα εγκρίνεται. Une abstention. Ah oui, une abstention. Ah, με μία αποχή. Εντάξει, για να μην του φουσκώσουν και τα μυαλά του κυρίου Μπέρμα, να έχει και μια αποχή. Δεύτερη γνωμοδότηση, πάλι ο μπλοκ ψηφίζουμε. Υπέρ των τριών τροπολογιών, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est εγκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια κύριε Μπέρμαν. Περνάμε στην έκθεση της κυρίας Σνίμπε Γιάστρα. Αρχίζουμε με την τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 2. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Για την παράγραφο 4. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται ψηφοφορία για την τροπολογία 7. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία... Α, ξέχασα την 8, συγγνώμη. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ξανακάνω την 9 για να μην μπερδευτούμε. 9 ξανά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Euh, λοιπόν, έκθεση Κάσμαν. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, γιατί 2 υπέρ, ξανά, κατά, Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε επαληθεύσουμε για την τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3, υπέρ. Α, καταπίπτει. 4, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Για να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Σήμερα είναι δύσκολο. Για την τροπολογία 4, λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 6. Καθυστερείτε νομίζω. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 7 καταπίπτει. Για την τροπολογία 2, προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία. Πέραση της ε, ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 8 καταπίπτει. Να ψηφίσουμε χωριστά. Άρα ε, δίκιο είχα, καταπίπτει. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά.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 καταπίπτει και 17 καταπίπτει, 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Ομόφωνα εγκρίνεται συγχαρητήρια. Κύριε Μπέρμαν, θέλετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω το εξή. Άμα ξενυχτήσετε στο αεροπλάνο, πρέπει να σας πω συγχαρητήρια, γιατί τα πάτε πολύ καλά, Πρόεδρε. Λοιπόν, και έχουμε φτάσει στην έκθεση Σβένσον. Il paraît que je vais trop vite. Τώρα μου λένε ότι τα λέω πολύ γρήγορα. Εγώ νόμιζα ότι δεν τα λέω γρήγορα σήμερα, λέει η πρόεδρο. Uh, Στην τροπολογία 32 κάτι έχουμε να πούμε, θα το πούμε όταν φτάσουμε εκεί. Ξεκινάμε με την τροπολογία 38 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, επαληθεύουμε. Για τη 41 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 43 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 σε δύο τμήματα υπέρ, του πρώτου τμήματος, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της 49. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στροπολογία 50 πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της στροπολογίας 50. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Όχι, στο δεύτερο τμήμα έχουμε μια προφορική τροπολογία. Ανάμεσα στα δύο τμήματα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα τώρα. Πήγα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, για ξανά. Προφορική τροπολογία. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 της ΙΝΤΑ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 και 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56. Καταπίπτει η 56. 57 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ωραία. Πέραση τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 5. συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Α, όχι, να επαληθεύσουμε. Την 64 επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά ε, επαληθεύουμε για την 67 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 5 της ΙΝΤΑ ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ίντα 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. τα 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. τα 8 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. τα 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τα 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τα 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τα 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τα 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτουν οι επόμενες και φτάνουμε στην 72. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση. Για την 74 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 σε δύο τμήματα. Με μια προφορική τροπολογία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Αλλά θέλω και λίγο ησυχία στην αίθουσα. 79 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση. Ναι, ναι. Υπάρχει ένσταση για την προφορική τροπολογία. Περνάμε στο δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υπάρχει και τρίτο τμήμα. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά. Να επαληθεύσουμε την τροπολογία 82, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ίντα 1, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε την 85. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 91, συγγνώμη, υπέρ, κατά. Επαληθεύουμε την 91, άρχεται η ψηφοφορία. Για την προφορική τροπολογία νομίζω ότι υπάρχει αντίρρηση. 92. Καταπίπτει ή όχι. Όχι, δεν καταπίπτει. 92 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. τα 2 υπέρ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 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και εγώ γιατί είχα πει ότι εγκρίθηκε. Α, 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 δύο τμήματα η πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 104 ηλεκτρονικός έναρξη ψηφοφορίας πέρας εγκρίνεται. τα 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108. 108 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές δεν ξέρω. Να ελέγξουμε. Νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά δεν είμαι σίγουρη. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 108. Πέρας. Εγκρίνεται. Καλά κάναμε και το ελέγξαμε. 109 δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. να το ελέγξουμε. Για την 110.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 Αποχές εγκρίνεται. 119 δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά.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 Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να την, να την ελέγξουμε την 15. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Κύριε Κάσμαν, ε, δεν κατάλαβα. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορία για τη 16. Πέρας. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικός έναρξη ψηφοφορίας. Είμαστε στη 18, λέει η πρόεδρο. Συγγνώμη, έχω κάνει λάθος. Στη 18 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά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 εγώ προσπαθούσα να ε, ενθαρρύνω την ε, φιλία μεταξύ των λαών. Είναι σημαντικό. 28 τροπολογία καταπίπτει. Να δούμε τι άλλο καταπίπτει. Φτάνουμε στην 31. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Δύο τμήματα. Αχα. Ποιο είναι το πρόβλημά μας εδώ χωρίς το by the EU. Λοιπόν, το πρώτο τμήμα είναι χωρίς τις λέξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, by the EU. Ψηφίζουμε την 32, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές, τι να σας πω, μπορείτε να είστε λίγο πιο πειθαρχημένοι, να την ελέγξουμε αυτήν, αφού το ελέγξουμε αυτό το πρώτο τμήμα. Άντε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, μα σηκώστε τα χεράκια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 Ηλεκτρονικό έλεγχο 34 έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. αργείτε. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.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 ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της έκθεσης, έναρξη ψηφοφορίας. Πολύ αργείται. Πέρασα. Εγκρίνεται. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Après, après, après. Euh, Να κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί είναι εδώ μια ομάδα διπλωματών από τη Σαουδική Αραβία ε, που θα μας κάνουν παρέα στην ψηφοφορία. Καλώς ήρθατε. Ωραία. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Τυρουλιά. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Οι άλλες καταπίπτουν. 14. Υπέρ. Κατά. Δεν γίνεται τίποτε. Ψηφίζουμε τη 14. On vote. Oui, on vote, on vote. C'est cette partie-là qui n'est pas. Ah. D'accord. Donc, il y a une partie. Υπάρχει ένα, πτυχίο, ένα στοιχείο γλωσσικό που δεν το ψηφίζουμε, αλλά ψηφίζουμε η τροπολογία 14. Οπότε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Δύο, δύο τμήματα. Υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτει επόμενη συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20-21 καταπίπτουν, προφορική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ. Κατά, α, καταπίπτει. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7 της Επιτροπής Προϋπολογισμών υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 κατά πίπτη. 27 υπέρ. Υπέρ. 27. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28. Καταπίπτει. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. τις 31. Πέρας. Απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ποιος λέει όχι. Κάποιος φωνάζει όχι. Et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 Μιλάω για την παράγραφο 16 και την ε, τροπολογία του κυρίου Πόγκα που είναι ξεχωριστή τροπολογία. Είναι τρία τμήματα και πρέπει να ξανακάνουμε αυτή την ψηφοφορία. Λοιπόν, άρα, τρία τμήματα του κυρίου Πόγκα λέω τώρα. Είναι ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία. Πάμε στην 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προφορική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Α, 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 τρία τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικό στο δεύτερο τμήμα της 37 έναρξη ψηφοφορίας πέρας εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 38. Κατέπεσε. 39 τότε υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος 39 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται προφορική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα τώρα πάμε στη συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το προπολογισμό, παράγραφος 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τον προϋπολογισμό παράγραφος 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία. Όχι, όχι, την 53 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται προφορική 10 υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Μπιτζ 2 υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μπιτζ 3 υπέρ, Μπορούμε να τα ψηφίσουμε όλα μαζί από, 3 μέχρι, από το 3 μέχρι το 10 των προπολογισμών. Ωραία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά. Φαμ. Ομπλοκ. Όχι. Παράγραφος 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά να κάνουμε συνολική ψηφοφορία από τις ΦΑΜ 2 μέχρι 18.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 έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, πέρας, υπέρ, εγκρίνεται. Λοιπόν, 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 19, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φαμ 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Προφορική τροπολογία 11 πόγκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προ... Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φαμ α. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. B. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται φαμ C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται E υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται F υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται G υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται H υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 εγκρίνεται. τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικός. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. C'est bon <laughs> Alors, nous allons continuer. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Κυρία Μάισνερ, η έκθεση κυρία Μάισνερ. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικός. Εντάξει, Πέρασα. Εγκρίνεται. Ησυχία. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Τυρολιά. 30. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16. Υπέρ κατά αποχές της αποσχόλησης. 17. Υπέρ κατά αποχές. 18. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ε, εμπλουά. 20. Υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική υπαριθμών 1. Υπέρ Ναι, 21. Ε, εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Έργατα αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία, τροπολογία, τροπολογία, η 22, απασχόλησης, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, συμβαστική β υπέρ κατά εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία συμβαστική σε υπέρ κατά εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Αελίας ε, 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 α όχι όχι γίνεται 11 συγγνώμη 11 11 π είναι υπέρ κατά εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απασχόλησης 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ εγκρίνεται 25 απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 27 απασχόληση υπέρ κατά ε, εγκρίνεται προφορική υπαριθμών 2 υπέρ κατά ε, εγκρίνεται 50, 28 ποια είναι 28 29 απασχόληση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απασχόληση 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απασχόλησης 31 σε δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρκατα εγκρίνεται, το δεύτερο υπέρκατα αποχές απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Απασχόλησης 32 υπέρκατα αποχές εγκρίνεται, απασχόλησης 33 σε τρία τμήματα. Το πρώτο πι υπέρ, πίνε κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Απόσχολες 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξαναρχίζω, ξαναρχίζω γιατί δεν τα είδα. Απασχόληση 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απασχόλησης. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απασχόληση 37 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απασχόληση 39 υπέρ κατά απόχέ, απορρίπτεται απασχόληση 40 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται απασχόληση 41 σε δύο τμήματα το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ ψήσουμε όλες μαζί από την 45 μέχρι το 56 ναι ωραία πάμε όχι όχι καλά ναι όλες μαζί από το 45 μέχρι το 56 είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται όλες μαζί από το 58 μέχρι το 52 όχι 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά από την αρχή για το 59 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά πέρας απορρίπτεται Πασχόλης 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Αποχές. Και εγκρίνεται. Από το 53 όλες μαζί μέχρι το μέχρι το 66. Όχι, όχι. Με το, άντε, μέχρι το 64. 84. 84. Πού είναι. Δεν υπάρχει. Propose du 53 au 58. 53 μέχρι 58 σας προτείνω. Είναι υπέρ το το 53 μέχρι το 58. Υπέρ κατά εγκρίνονται από την 60 μέχρι την 66. Ναι, ναι, ναι, όλες μαζί. Non, c'est pas possible. Donc, je... Αδύνατο, αδύνατο. Επομένως σας προτείνω να ψηφίσουμε. Ακούστε, ακούστε. Προτείνω από το 60 μέχρι τη συμβαστική δέλτα. Οκ. Okay. Καλώς. Υπέρ κατά εγκρίνονται. 68 ε, υπερκατά εγκρίνονται. 17 ε, υπερκατά αποχές εγκρίνεται. 16 ήταν πριν, συγγνώμη, 16. Το 17 και εγκρίνεται και αυτή. Τώρα το 18 μέχρι το 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σας προτείνω όλες μαζί από το 21 μέχρι το 84. Καλώς. Υπέρ κατά εποχές εγκρίνονται. Ε, καλά, αυτό εγώ το ερμηνεύω ως άρνηση. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές παραγράφους. Υπερθυμών 1 εγκρίνεται. Ε, Απασχόλησης 1 υπερκατά εποχές εγκρίνεται. 2 απασχόληση υπερκατά εποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται. Προσκοπησίες 3 υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται. Όλες μαζί από την απασχόληση 4. Α, όχι, όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Απασχόλησης 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. αποσχολήσει 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 ε, σε τρία τμήματα υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω το αποτέλεσμα, δεν είναι σαφές, ξαναψηφίζουμε ε, ηλεκτρονικά για το πρώτο τμήμα της 11. Πέρα δεν εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12, από το 12 μέχρι το 14 μαζί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται απασχόλησης 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται τροπολογία εγκρίθηκε, ναι, ναι εγκρίθηκε άρα πάμε στο 29 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφορία ψηφίζουμε Ορισμένοι από εσά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγκρίνεται ομόφωνα, συγχαρητήρια. Τι θα πρέπει να ξαναψηφίσουμε, τι ψηφίσαμε δύο φορέ. Il faut également voter sur la résolution. Θα πρέπει να ψηφίσουμε και το σύνολο του ψηφίσματο. Το νομοθετικό ψήφισμα. Ψηφίζουμε.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 Alors, avant Πριν συνεχίζουμε, θα πρέπει να καλωσορίσουμε μια ομάδα επισκεπτών από την Τουλούζη. Τους ε, κάλεσε η κυρία Γκρέζ για τους πράσινους. Καλωσορίσατε. Θα συνεχίσουμε τώρα. Έκθεση Λέβιν. Τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές επαλήθευση. Le Και απορρίπτεται. Προφημόν ένα προφορική υπερκατάποχες εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Κάποιοι καθυστερούν. Mm. Πέρας. κρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Λέβιν. Η τελευταία ψηφοφορία. Έκθεση Ζαμπόρσκα. Alors, le dernier, Madame Zaborska, nous a τελευταία τη κυρία Ζαμπόρκα και αρχίζουμε από την παράγραφο 1. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ, κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά. Αποχέ. Ελεκτρονική ψηφορία για επαλήθευση για το 2. Ψηφίζουμε. Α, πάτε πιο αργά από Πολύ καλά. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1, η 2, υπερκατά εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 1, υπερκατά αποχές, εγκρίνεται. 6, υπερ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομοφόνο. Συγχαρητήρια κυρία Ζαμπόσκα. Merci. Alors, vous n'êtes pas obligés de partir, hein, messieurs les députés. Messieurs et mesdames les députés, vous n'êtes vraiment pas obligés de partir. Όχι, όχι, όχι, δεν πρέπει να αποχωρήσετε, κύριοι συνάδελφοι.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 Sì, sì, sì, sì, sì, sì, ah, offre il tuyo. Ok, ok, entonces, te, te arreglo ahí entonces. Nous allons continuer. Θα συνεχίσουμε. Αυτοί που θέλουν κοβεντούλα μπορούν να αποχωρήσουν. Nous passons maintenant à la... Τώρα. Πάμε στην παρουσίαση του ενημερωτικού εγγράφου σχετικά με την επισκόπηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη φτώχεια mm Mm-hmm ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για καταπολέμηση διακρίσεων λόγω κοινωνική τάξη. Έχουμε μια σειρά από ψηφίσματα που αφορούν ε, αυτό το πρόβλημα ε, για τις κοινωνικέ τάξεις και το 2007, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Το 2011 θέλουμε να οργανώσουμε με την Υποπιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα μια ακρόαση όσον αφορά τι δυσμενεί διακρίσεις λόγω κοινωνική τάξη στην Νότια Ασία. το λόγο ε, στους εισηγητές θα πρέπει να σας πω κάποιες ιδέες. Θα ήθελα να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου ε, οι διακρίσεις λόγω και κοινωνικής τάξης είναι πιο σοβαρές σε με τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι μία από τις πιο δεδομένες διακρίσεις γιατί έχουμε πάνω από 200 ε, εκατομμύρια οι οποίοι είναι θύματα και κυρίως αυτοί που γενικούν στην Νότια Ασία ε, καταπολέμηση των δικαιωμάτων τους, των πιο θεμελιωδών και είναι βασικές πρακτικές που γίνονται και να μπορούν να έχουν προσβασιμότητα στις βασικές δημόσιες υπηρεσίες, να μην έχουν δουλειά, και οπότε έχουμε και τέτοιες άλλες διακρίσεις κοινωνικής τάξης. Θέλω να πω τελευταίο ότι είναι μία από τις βασικές αιτίες για τη φτώχεια και αυτό είναι ένα εμπόδιο όσον αφορά τους στόχους του, του, του, του, 2000 ε, και τώρα θα δώσουμε το λόγο στους ε, ειδικού, του εμπειρογνωμονέ μα και θα ξεκινάμε με την κυρία Λάγκσδορφ και κατόπιν οι υπόλοιποι. Ξεκινούμε δίνοντα το λόγο στου εμπειρογνώμονε που θα μα παρουσιάσουν αυτή τη μελέτη. Και θα ξεκινήσουμε, ναι, τελικά με την κυρία Λάγκσδορφ, η οποία εργάζεται για το Οικολογικό Ίδρυμα. Ε, έχετε maximum 10 λεπτά. Έχετε το λόγο, κυρία. Okay. <clears throat> Thank you very much. Um, Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αναθεώρηση σχετικά με τη φτώχεια. Διακριτική μεταχείριση με βάση την ε, κοινωνική τάξη. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο και γι' αυτό θα ε, πω δυο εισαγωγικά λόγια και στο δεύτερο τμήμα θα μιλήσω για την διακριτική μεταχείριση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα μιλήσω για τη διακριτική μεταχείριση, τον τύπο διακριτικής μεταχείρισης και το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πέντε συγκεκριμένες χώρες, Μπαγκλαντές, Ινδία, Νεπάλ, Πακιστάν και Ιεμένη. Και τέλος, ε, κάποια από τα συμπεράσματα και τις συστάσεις τα οποία έχουμε καταλήξει και το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει τη διακριτική μεταχείριση με βάση την κοινωνική τάξη σε αυτέ τι χώρε και σε άλλε. Νομίζω ότι όλοι έχουν κάποια εικόνα του τι είναι οι κάστε, οι κοινωνικέ τάξει. Οι κάστε ε, έχουν μια κοινωνική διαστρωμάτωση, διαχωρίζονται οι ομάδε με κληρονομικό διαχωρισμό εργασία, έχουν σχέση με τον Ινδουισμό, αλλά περισσότερο είναι οργανωμένε με βάση τα επαγγέλματα, δηλαδή δεν υπάρχουν μόνο Στι χώρε τη νότια Ασία, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου, στην Αφρική παραδείγματος χάρη και στην Ιαπωνία και στο Μπαλί. 260 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο πλήττονται από αυτή τη διακριτική μεταχείριση. Από αυτούς 167 ε, εκατομμύρια ζουν στην Ινδία και υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Νότιας Ασίας ε, και αλλού όπως σας είπα. Η Dalit είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Είναι έξω από το παραδοσιακό σύστημα με τις κάστες γιατί δεν ε, εντάσσονται σε αυτή, σε αυτή την κατηγορία. Πριν ε, δημιουργηθεί η χώρα, δημιουργηθεί η το 1949, ονομάζονταν παρίες και συνεχίζει αυτή η πρακτική με τους παρίες σε πολλά τμήματα της χώρας. Περισσότερο πλήττονται οι γυναίκες και με βάση όλους τους δείκτες οι γυναίκες βρίσκονται στο πιο χαμηλό, στη πιο χαμηλή στάθμη όσον αφορά την εκπαίδευση, τον ευάλωτο χαρακτήρα, τη δυνατότητα να υπερασπίσουν τον εαυτό τους και υπόκεινται σε βία και σε σεξουαλική βία. Είναι ένα είδος υποκατηγορίας ε, και τους ανατίθεται δουλειά που τις υποβαθμίζει, παραδείγματος χάρη να ψάχνουν στα σκουπίδια. Άλλη ευάλωτη ομάδα είναι ε, τα παιδιά, διότι δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και αυτό είναι μια σοβαρή διακριτική μεταχείριση. Όπως ήδη είπαμε, βλέπω ότι δεν έχουμε καθόλου χρόνο και πρέπει να βιαστώ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η βία, που μπορεί να είναι σωματική ή ηλεκτρική βία, ε, το ότι δεν τους δίδονται δικαιώματα, περιορισμοί στην κοινωνική και θρησκευτική ζωή, δεν τους επιτρέπουν την είσοδο σε ναούς, παραδείγματος χάρη, ή δεν μπορούν να θάψουν τους ε, ναούς τους ή να χρησιμοποιήσουν ε, δημόσιες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης. Δεν έχουν πρόσβαση σε πόρους και υπηρεσίες. Υφίστανται ένα κοινωνικό και οικονομικό μποϊκοτάζ. Όσον αφορά την απασχόληση, όπω σα είπα, είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα, γιατί οι κάστε είναι οργανωμένε με βάση την απασχόληση. Ορισμένε λοιπόν δουλειέ που θεωρούνται ακάθαρτες είναι δουλειέ που δίδονται στι χαμηλέ τάξει και στους ντάλιτ. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη επίσης είναι ένα πρόβλημα και συμμετοχή στα πολιτικά ζητήματα. Υπάρχει νομοθεσία συνήθως, αλλά η εφαρμογή της νομοθεσίας δεν γίνεται με επαρκή τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει προσπαθήσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα της διακριτικής μεταχείρισης με βάση την κοινωνική τάξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάποια ψηφίσματα τα οποία έχουμε παραθέσει σε αυτό τον κατάλογο, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Τάλι στην Ινδία ε, το 2012, και άλλα παλαιότερα ψηφίσματα. Εδώ υπήρχαν δύο άρθρα για την διακριτική μεταχείριση με βάση την κοινωνική τάξη και για την Ινδία συγκεκριμένα. όπου αντιμετωπίζονται και κάποια από τα πιο σοβαρά προβλήματα. Έχουν γίνει και πολλές ακροάσεις, ε, συνεχίζεται η αναπτυξιακή συνεργασία, αλλά ακόμη δεν έχει συμπεριληφθεί το θέμα στην ετήσια έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι διάβλους βοηθείας έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν, ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αναπτυξιακή συνεργασία, η ανθρωπιστική βοήθεια και οι εμπορικές σχέσεις. Τώρα θα περάσω στο επόμενο μέρος της παρουσίασής μου για το πώς ε, ε, έχουμε αντιμετωπίσει το θέμα σε πέντε χώρες. Ξεκινώ με τον Μπαγκλαντές για να σας δείξω ότι είναι σημαντικό και σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο περιφέρειας να γίνεται η δουλειά και τονίζω το ότι χρειάζεται ενημέρωση και πληροφόρηση στο Μπαγκλαντές Απαντάτε η διακριτική μεταχείριση με τις μορφές που σας προανέφερα. Διαχωρισμός, διακριτική μεταχείριση με βάση ε, ε, ε, την κοινωνική τάξη όσον αφορά την απασχόληση. και συνήθως δεν υπάρχει επίγνωση μεταξύ των ίδιων των ε, πολιτών αυτής της κοινωνικής ε, τάξης για τα δικαιώματά τους ε, και έχουν χαμηλή πολιτική εκπροσώπηση. Μπορεί να υπάρχει το νομικό πλαίσιο, αλλά δεν έχουν οι την επίγνωση των νομικών τους δικαιωμάτων. Ε, και ε, στη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μπαγκλαντές έμφαση δίνεται στην αναπτυξιακή συνεργασία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μια προτεραιότητα και δεν έχει τεθεί έμφαση στην διακριτική μεταχείριση με βάση την κοινωνική τάξη. Δεύτερο παράδειγμα, η Ινδία. Η Ινδία έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό Dalit και άλλων χαμηλών κοινωνικών τάξεων και επίσης ε, έχει διαφορετική βαρύτητα σε σχέση με τις άλλες χώρες η Ινδία. Τα θέματα της διακριτικής μεταχείρισης με βάση τις κάστες έχουν συζητηθεί τα τελε... Ε, ε, μεγάλο αριθμό ετών. Είπαμε ότι ανατίθενται ταπεινωτικέ δουλειέ σε αυτέ ε, τι κατηγορίε πολιτών, παραδείγματο χάρη ο καθαρισμό αποχωρητηρίων με τα χέρια. Και παρότι υπάρχει το νομικό πλαίσιο για τους παρείες ε, ήδη από το Σύνταγμα του 1949, συνεχίζουν να υπάρχουν ε, κάποιες ποσοστώσεις για τους Ντάλιτ. Η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη παραμένει σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Στην Ινδία είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα αυτό και είναι δύσκολο να το θίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρεται σε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει στις διασκέψει κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδίας να συζητηθεί αυτό το θέμα, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη αυτό. Στις τρει τελευταίες διασκέψει κορυφής Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδίας δεν έχει αναφερθεί και στα πιο σημαντικά έγγραφα θα έπρεπε να αναφέρεται. Όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία, έχει συμπεριληφθεί το θέμα της διακριτικής μεταχείρισης, αλλά όχι με τρόπο συνεπή και συνεκτικό εξετάσαμε και κάποια συγκεκριμένα αναπτυξιακά προγράμματα όπου βλέπουμε ότι μερικές φορές θίγεται το θέμα αλλά όχι με συνέπεια. Επόμενο παράδειγμα, το Νεπάλ. Στο Νεπάλ έχει γίνει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης με βάση την κοινωνική τάξη. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν γίνει πολλά βήματα Απαγορεύτηκε η διακριτική μεταχείριση το 1990. Το 2009 αποφασίστηκε ότι θα εκλείψει ε, η διακριτική μεταχείριση και το 2011 ψηφίστηκε και ένας νόμος σχετικά με τους παρείες και τη διακριτική μεταχείριση με βάση την κοινωνική τάξη. Εποφελήθηκε λοιπόν τον Νεπάλ σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει δουλέψει πολύ και με τα Ηνωμένα Έθνη και με τις σχετικές συστάσεις. Περνώ στο Πακιστάν και στην Ιεμένη. Είναι άλλα δύο παραδείγματα που συνήθως δεν τα συνδυάζουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για αυτό το θέμα. Υπάρχουν μεγάλες ομάδες Dalit και χαμηλών κοινωνικών τάξεων και στις δύο αυτές χώρες, αλλά δεν υπάρχει αναγνώριση του προβλήματος και επίγνωση μέσα στην κάθε χώρα και γι' αυτό δεν εντοπίζεται και στις συμφωνίες συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλήγω τέλος στα συμπεράσματά μας και στις συστάσεις μας. Το πιο σημαντικό είναι ότι σε οποιαδήποτε αξιολόγηση θα πρέπει να ληφθούν ε, υπόψη αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί για τις κοινωνικές τάξεις, διότι πολλές τέτοιες κοινωνικές τάξεις υφίστανται διακριτική μεταχείριση. και θα πρέπει να συγκεντρωθούν πληροφορίες τις οποίες ε, να μπορούν ε, στις οποίες να μπορούν να έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι. Από ε, τον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουμε πάρει πολλά διδάγματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σε αυτή την περίπτωση των ε, διακριτικών μεταγυρίσεων με βάση την κοινωνική τάξη και σε βασικούς τομείς όπως είναι η εκπαίδευση και η δικαιοσύνη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτό το θέμα της κοινωνικής τάξης. Θα πρέπει να γίνεται με ελάχιστες συστάσεις για αυτούς τους τομείς που θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Μετά το τσουνάμι συγκεκριμένα, οι μελέτες που έγιναν έχουν δείξει ότι τα μέλη χαμηλών κοινωνικών τάξεων ήταν ιδιαίτερα ευάλωτα και δεν λάμβαναν και την ε, βοήθεια που ε, παρεσχέθη μετά τη φυσική καταστροφή. Πρέπει λοιπόν και στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην αναπτυξιακή συνεργασία να ληφθεί υπόψη αυτό το πρόβλημα της διακριτικής μεταχείρισης ε, για να μπορούν και να ενημερωθούν ε, οι ενδιαφερόμενοι και να δίνεται πληροφόρηση και στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με αυτές τις υποθέσεις έχει συγκεντρωθεί ένας όγκος γνώσης για τους Ντάλιτ και τις χαμηλές κοινωνικές τάξεις και θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κάποια σημεία επαφής που συγκεντρώνουν ε, αυτό τον πλούτο πληροφοριών για τις κοινωνικές τάξεις και τους Ντάλιτ. Λοιπόν, αυτές είναι κάποιες ε, Αυτά είναι κάποια στοιχεία που μπορείτε να λάβετε υπόψη σας. Ζητώ συγγνώμη, λέει πρόεδρο που σας διακόπτω, αλλά ήδη έχουμε πάρει χρόνο από, τη, από τις επόμενες παρουσιάσεις. Και δίνω το λόγο στο δίκτυο ελληνικής για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστούμε που μας ε, δίνει την ευκαιρία να συνεισφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Το ώστε να σταματήσει αυτού του είδου η δυσμενή διάκριση, γιατί όπως είπατε έχει να κάνει με 260 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο και περισσότεροι εξ αυτών ζουν στην Ανατολική Ασία. Οι περισσότεροι από αυτούς, τους ντάλιτς ή τους λεγόμενους άθικτους, η ε, διεθνής διάκριση σημαίνει φτώχεια, ταπείνωση. Δεν έχουν τα βασικά δικαιώματα, δεν έχουν τη βασική αξιοπρέπεια ως άνθρωποι παρά το Σύνταγμα, κάποια μέτρα και κάποια νομοθετήματα ε, στις χώρες όπου ξοδεί αυτό το φαινόμενο. Ε, αυτού του είδου η διάκριση είναι συνεχές φαινόμενο και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν προσβασιμότητα στις βασικές υπηρεσίες, σχολείο, νερό, στην αγορά, στην απασχόληση και επίσης στις περισσότερες ε, περιπτώσεις ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας, ε, βέβαια συνδέονται με αυτή τη μορφή και άλλες μορφές διάκρισης, Οπότε έτσι έχουμε σώρευση αυτού του φαινομένου, είναι πιο ευάλωτοι αυτοί οι άνθρωποι και κυρίως ε, οι ανήλικοι και οι γυναίκες αυτής της κοινωνικής τάξης. Ε, εξαναγκαστική εργασία, ε, κακοποίηση, βασανιστήρια, οπότε επομένω πρόκειται για ε, δομικό στοιχείο της φτώχειας, της του κοινωνικού αποκλεισμού, οπότε τέτοιου είδους δυσμενής διάκριση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με συστηματικό τρόπο και με πολυμερή μέθοδο στα πλαίσια του προγράμματος για το 2015 στα πλαίσια της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημείωσε και τόνισε με το ψήφισμα του, του, του Δεκεμβρίου, έχουμε στοχευμένη ε, βία κατά των γυναικών, κατά των αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως στην Ινδία αλλά και σε άλλες χώρες. Όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια της γενικότερης ε, αποτυχίας του να εφαρμοστεί ο και πολλές φορές ε, έχουμε στις χώρες αυτές που δεν λειτουργούν τα δικαιώματα πάρα πολλές σοβαρές παραβιάσεις και έχουμε ε, κάποιο είδους ε, συνθήκες, συμβάσεις, αναθεώρηση νομοθεσίας. Παρ' όλα αυτά όμως συνεχώς έχουμε όλο ένα και περισσότερη παραβίαση των δικαιωμάτων λόγω κοινωνικής τάξης και παρά τις συστάσεις προς τη, τις κυβερνήσεις και τα διαφθασμικά όργανα και επομένως ο ΙΕ έχει προμαστεί γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι ε, πάρα πολύ βασική υπόθεση για να υπερτανεύσει τελικά η ισότητα να αποκλειστούν οι διακρίσεις και γι' αυτό και καλούνται τα μέλη του ΟΗΕ να αναλάβουν δράση στο Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και κυρίως έτσι να υπάρξει ένα πλαίσιο για να σταματήσει σταματήσουν αυτού του είδου δυσμενείς διακρίσεις. Οπότε, με αυτά υπόψη και λαμβάνοντα υπόψη το τι έχει κάνει το Ευρωκοινοβούλιο και την σύσταση που έχει διατυπώσει, συνεχίζουν να μένουν αναπάντητα κάποια ερωτήματα και δεν έχει δοθεί συνέχεια σε εκείνη τη σύσταση του Κοινοβουλίου. Άρα, επήγει να δοθεί νέα όθηση στο θέμα, σε διεθνή κλίμακα, να προβληθεί το θέμα και να το δοθεί υψηλή προτεραιότητα. Είναι πρόβλημα ανάπτυξης, είναι πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε και να υπάρξει η βάση για ένα επικοδομητικό διάλογο για τις φυγόμενες χώρες. Θα πρέπει βέβαια να υποστηριχθεί οικονομικά αυτή η προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται του Ντάλιτ μια στήριξη βέβαια, αλλά χρειάζεται και μια προσέγγιση που να περιλαμβάνει ε, σφαιρικότητα που να είναι, έχει σφαιρικό χαρακτήρα συνολικό. Και προτείνουμε λόγω της κλίμακας του μεγέθους του προβλήματος η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει πιο συστηματικά, πιο μεθοδικά σε όλες τις, τις πολιτικές αυτό το πρόβλημα και στις συμφωνίες σύνδεσης και στα προγράμματα. Έχει δείξει εμπειρία ότι όταν δεν μπορέσουμε να ξεπεράσουμε συγκεκριμένε τέτοιε προκλήσει σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι κοινωνικέ τάξει, έχουμε ε, έλλειψη στρατηγικών δεδομένων, ε, ε, ανάλυση πολιτικής, κατάλληλα εργαλεία. Έχει όμως τα εργαλεία, έχει τα μέσα στη διάθεση της Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε ένα σωρό θετικές, Προτάσει σε αυτή τη ε, μελέτη για το τι θα μπορούσε να γίνει, καθημερινέ γραμμέ, προγραμματισμό σε κρατικό επίπεδο. Οπότε είναι σημαντικό όλα αυτά να καλυφθούν από τι στρατηγικέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να, να περισσότερο το θέμα στον διάλογο των ανθρώπινων δικαιώματα. Ολοκληρώνουμε τρία βασικά σημεία, μια σφαιρική, πολιτική για αυτό το πρόβλημα αυτό, συστηματική προσέγγιση με ό,τι μέσα έχει στη διάθεσή τη να το αντιμετωπίσει αυτό. Οι πολιτικέ, στρατηγικέ, προγράμματα δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσα να σα δώσω παραδείγματα, αν δεν έχουμε το χρόνο, ε, αναπτυξιακή βοήθεια, ανθρωπιστική αρρωγή, ε, εμπόριο, επιχειρηματικότητα και θα πρέπει επομένω να γνωριστεί το φαινόμενο αυτή τη διάκριση και επομένως θα πρέπει να του δοθεί δέουσα προσοχή με εγκάρσιο τρόπο σε όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πιο ενεργή πολιτική, πιο συστηματική πολιτική για τον και τον διάλογο και να χρησιμοποιηθούν όλες οι στάσεις του ΟΗΕ που υπάρχουν, που είναι δεδομένες και εν κατακλείδη θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλέξει περισσότερο την κοινωνία, να έχει πιο δυναμική προσέγγιση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σε επίπεδο ΟΗΕ από πλευρά των, των μελών ε, κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδείχνει το θέμα. Κάποιε αρχέ, κάποιε καθημερινέ γραμμέ και. Σα ευχαριστούμε, ευχαριστούμε λοιπόν. Μισό, μισό, μία φράση, μία φράση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα ως κάποια διάκριση ε, και να θεωρηθεί το ίδιο σημαντική όπως οι άλλες διακρίσεις με τη βάση του φύλου και λοιπά και βάση των γενετησίων ε, προτιμήσεων και λοιπά. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους ευρωβουλευτές. Σας το λέω, είμαστε πολύ καθυστερημένοι και θα θέλα να σας ζητήσω να είστε σύντομοι. Ο κύριος Ντάνσκης. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπατε σε σχέση με τις διακρίσεις λόγω κάστα, λόγω κοινωνική τάξη, το να προσπαθείτε τώρα να το συνδυέσετε ε, με το φύλλο ε, είναι δύσκολο γιατί πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιούμε τον πολιτιστικό σχετικισμό για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε κάτι τέτοιο, τέτοιου είδους διακρίσεις, λόγω δηλαδή της μοναδικότητας ενό, ενός πολιτισμού. Έτσι το δικαιολογούμε δηλαδή, το οποίο πραγματικά είναι μια σκανδαλώδης ανοησία. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ε, ασχοληθεί με αυτό το θέμα των ανέγγιχτων, των Ντάλιτς, ε, να υπάρχει δηλαδή μια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Προσπαθούμε, πρέπει να προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο μέσο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και συμφωνώ με την έκθεση πρωτοβουλία, θα την υποστηρίξω απολύτω την έκθεση πρωτοβουλία ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Δίνω το λόγο στον κύριο Κάσμαν, λέει πρόεδρο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Νόλου και την κυρία Λάγκστορφ για τις παρουσιάσεις τους και συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπε ο κύριος Δόνσκης. Ε, ε, είναι αυτό που λέγαμε χθε σε σχέση με τις διακρίσεις ε, που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ε, ή οι άνθρωποι λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Πάντοτε η δικαιολογία είναι ο πολιτισμός. Ε, όχι, τότε ο πολιτισμός πρέπει να αλλάξει, πρέπει να εξελιχθεί. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα, είναι εγκάρσια, επηρεάζει το θέμα αυτό πολλές ε, επιτροπές ε, στο κοινοβούλιο μας και συμφωνώ απολύτως με την ε, προσέγγιση αυτή. Πρέπει όμως να περάσουμε στην πράξη, να μετουσιωθεί σε πράξη μέσω έκθεσης πρωτοβουλίες από την Επιτροπή μας με ένα σχέδιο δράσης και ένα χρονοδιάγραμμα γιατί αυτό έχει άμεση σχέση με όλες τις υπόλοιπες μορφές διακρίσεων. Ευχαριστώ. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέζ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τις ε, δύο μιλήτριες ε, γιατί ήταν πάρα πολύ σαφής ε, και εκπαιδευτική η παρουσίαση τους. Έχω ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον να γνωρίζω τι μέθοδο, τι στρατηγική ε, εφαρμόζει η Επιτροπή, ώστε η διμερής βοήθεια η αναπτυξιακή από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρες όπου υπάρχει το σύστημα της κάστας ε, να ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση των διακρίσεων και κυρίως για την καταπολέμηση της ένδυας μεταξύ των ομάδων που πλήττονται από αυτήν τη διάκριση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ λέει η Πρόεδρος. Ναι παρακαλώ θα πάρω καφέ. Κύριε Μπέρμαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τις ομιλήτρες για αυτές τις δύο πολύ σαφείς παρουσιάσεις το πρόβλημα του πολιτικού διαλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με χώρες οποίες, ε, όπου υπάρχουν διακρίσεις λόγω καστών ε, είναι ακόμη δυσκολότερο στην, στην Ινδία γιατί είναι μια, ένα, μια, ισχυρό κράτος το οποίο δεν θέλει καν να ακούσει τέτοιου είδους κριτική. Λέει ότι η νομοθεσία μας είναι τέλεια, οπότε τι είναι αυτά που μας λέτε. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα παγκοσμιούμενο κόσμο με περισσότερους δωρητές από ό,τι στο παρελθόν στην αψυχική βοήθεια, από τους ιδιώτες ε, του Ιδρύματος του Bill Gates ε, ε, μεταξύ άλλων, πρέπει να προασπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες, τα ίσα δικαιώματα για κάθε πολίτη, οποιασδήποτε προέλευσης και οποιοδήποτε, οποιοδήποτε προσανατολισμού, ε, σεξουαλικού ή άλλου. Ο διάλογος είναι δύσκολος, αλλά είναι και καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα. Μία διόρθωση μόνο θα ήθελα να κάνω σε σχέση με την ε, έκθεσή σας για την, για την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των καστών, παρά το γεγονός ότι στο επόμενο αναπτυξιακό μέσο δεν θα υπάρξει δημαρής ε, βοήθεια προς την Ινδία, θα υπάρχει δυνατότητα στο πλαίσιο των θεματικών προγραμμάτων χρηματοδότησης της ενίσχυσης κοινωνίας των πολιτών και των σχετικών οργανώσεων στην Ινδία. Και είμαι πεπισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί να υποστηρίξει ειδικότερα ε, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, των Dalit, για να μπορέσουν και σε εθνικό επίπεδο ε, να ε, δουν τα δικαιώματά τους, να την χάνουν σεβασμού και προστασίας όπως θα έπρεπε. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Κύριος Κορτές Λάστρα. Πρώτα πρώτα Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τις δύο εμπειρογνώμονες που μας έκαναν τις εισηγήσεις τους Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι τελικά οι κοινωνικέ τάξεις έχουν να κάνουν με την κοινωνική διαστρωμάτωση. Και αυτό σχετίζεται και με το θέμα τη θρησκεία, με όλο το σεβασμό προ τι θρησκείε, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για πρόβλημα το οποίο αφορά εκατοντάδε εκατομμυρίων. Και βέβαια υπάρχει και μεγάλη δυσκολία για να να ξεφύγει από αυτό το σύστημα, από την κάθε κάστα, την κάθε κοινωνική τάξη δεν μπορούν, τους αρνούνται κάθε ανθρώπινο δικαίωμα για τον απλούστατο λόγο ότι ανήκουν σε μια κάστα και επομένω αναγκάζονται να συνεχίσουν να ανήκουν σε αυτή την κάστα και ούτω καταξής. Άρα το θέμα είναι θέμα παιδείας και βέβαια βρισκόμαστε τώρα ενώπιον ενός αδιεξόδου. Και αυτό νομίζω ότι είναι η ουσία, η διαστρωμάτωση ε, που δημιούργησε αυτές τις κάστες και είναι θέμα θρησκείας. Εμείς επομένως θα πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτό το πρόβλημα, ε, να το θεωρήσουμε δικό μας, θα πρέπει να προωθήσουμε ό,τι μπορούμε ε, με τη δουλειά εδώ στην Επιτροπή και μέσω του ΟΗΕ και ούτως ώστε να γίνει κάτι για την κοινωνία των πολιτών και με αυτήν. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σβένσον. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι είναι κρίμα που δεν έχουμε αρκετό χρόνο, χωρίς να παραπονούμε τώρα έναντι της Προέδρου, αλλά είναι κρίμα που δεν έχουμε χρόνο γιατί καλέσαμε προσκεκλημένους και δεν τους αφήσαμε χρόνο και έχουν την αίσθηση ότι τους διώχνουμε, ενώ για τέτοια θέματα θα έπρεπε να αφήνουμε πιο πολύ χρόνο γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Όταν μιλάμε για διακριτική μεταχείριση, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη διακριτική μεταχείριση με βάση την κοινωνική τάξη, όπως αυτό που λέμε τώρα για τις κάστες. Και θα θέλαμε από τους εμπειρογνώμονες που έρχονται ως προσκεκλημένοι να μας δώσουν ιδέες για να μπορέσουμε να τις έχουμε υπόψη μας. Δεν υπάρχει μόνο αυτός ο τομέας της διακριτικής μεταχείρισης όταν μιλάμε για τους Dalit. Παρότι δεν έχουμε εμείς κάποια λύση να σας δώσουμε σήμερα, ξέρουμε ότι είναι σημαντικό να γίνει κάτι για αυτά τα 260 εκατομμύρια πολιτών. Διότι πολύ συχνά μιλάμε για την Ευρώπη και για τη δημοκρατία. Όντως, η Ευρώπη είναι μια δημοκρατία που όμως δεν τολμά να μιλήσει για τέτοια προβλήματα. Και είναι κρίμα. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Όντω ο χρόνο πάντοτε μα πιέζει. Τι να κάνω, μα πήραν οι ψηφοφορίες πιο πολύ χρόνο, παρότι πήγα γρήγορα όσο μπορούσα. Τι να πω, πρέπει να βρούμε κάποιο σύστημα, γιατί όλα τα θέματα πάντοτε είναι σημαντικά. Και απογοητευόμαστε όταν δεν έχουμε αρκετό χρόνο για κάθε θέμα. Εμένα μου δίνουν χρόνο, προσπαθώ να τον τηρήσω, τι άλλο να κάνω. Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Λάγκστορφ καταρχήν για να απαντήσει, αν θέλει να απαντήσει σε κάποια σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα σας τα σχόλια. Σημείωσα μία ερώτηση που δεν απευθυνόταν καν σε μένα. Δεν ξέρω αν έχω να απαντήσω σε κάτι. Πάντως μετά από όλα τα σχόλια αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι όλοι συμφωνούμε Φαίνεται δηλαδή να είναι εύκολο αυτό το θέμα. Από την άλλη μεριά όμως είναι και πολύ δύσκολο, γιατί παρότι όλοι συμφωνούν είναι δύσκολο να κάνουμε κάτι. Και για την Ινδία όπως ελέγχθη. Έχουμε εντοπίσει κάποια σημεία όπου μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχουμε κάποιες ιδέες. Και σίγουρα θα προκύψουν και άλλες ιδέες, αρκεί να αφιερώσουμε χρόνο για να το συζητήσουμε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διδαχθεί πολλά από αυτά που έχει κάνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα. Πολλά από αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για την ε, διακριτική μεταχείριση με βάση τις κάστες. Αν δηλαδή χρησιμοποιήσουμε μια προσέγγιση όπου το θέμα αυτό θα περάσει σε όλες τις πολιτικές που χρησιμοποιούνται ε, ε, και εφαρμόζονται σε αυτούς τους τομείς, θα είναι χρήσιμο. Να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλει να παρέμβει. Ευχαριστώ. Μάρθα Μέντες Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν για την παρουσίαση της έκθεσης. Και ευχαριστώ και για την ε, ε, παρέμβαση της ομιλήτριας που έχουμε συναντήσει σε πολλές συνεδριάσεις μέχρι τώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των διαλόγων, του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ άλλων, και μέσω της θεματικής ε, υποστήριξης με χρηματοδοτικά μέσα σε συγκεκριμένες θεματικές ε, κάνει συγκεκριμένα βήματα για να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Και υπάρχουν παραδείγματα σε ορισμένες από τις χώρες αυτές παραδείγματα πρακτικών προγραμμάτων που λειτουργούν και που υποστηρίζουν τις χαμηλές αυτές τάξεις και που δίνουν τη δυνατότητα στους Ντάλιτ να βελτιώσουν τη θέση τους. Το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα βοηθά τους συναδέλφους στις αντιπροσωπείες να δουλέψουν με προγράμματα επιτόπου. Στις συζητήσεις για τα χρηματοδοτικά μέσα της επόμενης περίοδου προσπαθούμε να αποδώσουμε τη δέουσα σημασία στο θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να προσφέρουμε αυτά τα μέσα στους συναδέλφους μας στις αντιπροσωπείες επιτόπου. Εδώ έχουμε μια σειρά συστάσεων που μπορούμε να τις συζητήσουμε και πάντοτε είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα διακριτικής μεταχείρισης κατά των γυναικών, κατά των παιδιών κλπ. Αλλά σίγουρα είναι κάτι πάνω στο οποίο προσπαθούμε σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν κάποια μέσα διαθέσιμα, κάποια τα συζητάμε, κάποια έχουν ήδη εγκριθεί και προσπαθούμε να τα συζητάμε αυτά τα θέματα ε, για την κοινωνία των πολιτών και να τα χρησιμοποιούμε στα μέσα που διαθέτουμε. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Cashman, une petite Κύριε Κάσμαν, να κάνουμε μια εξαίρεση, μια και θέλετε το λόγο. Καλώς είναι σας, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. άκουσα την Επιτροπή που είπε ότι υπάρχουν κάποιες δράσεις. Φοβάμαι ότι έχουν αποτύχει αν υπάρχουν τέτοιες δράσεις της Επιτροπής. Άμα λέμε 260 εκατομμύρια πολίτες σε αυτές τις κατηγορίες, τι άλλο να πούμε. Και οι πράσινοι το έχουν θίξει αυτό το θέμα και μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας και θα ήθελα να σας ζητήσω να τεθεί ω θέμα στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών. Γιατί εδώ νομίζω ότι το Κοινοβούλιο έχει να κάνει κάτι. Très bien. Καλώς, λέει πρόεδρος. Καλώς. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε στο σημείο το οποίο αφορά την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σαχέλ. Μια μικρή αλλαγή είναι αυτή, διότι ο κύριος ε, Ποπόφσκι δεν έχει όμως ακόμα φτάσει δυστυχώς. Αλλά τέλος πάντων να ξεκινήσουμε για το Σαχέλ. Μια ε, περιοχή που έχει πάρα πολύ θυγή από κάποια προβλήματα που σοβούν εκεί, καταστροφές και βέβαια το βασικό θέμα αφορά εδώ πέρα την αδυναμία της διακυβέρνησης, τη φτώχεια και πρόκειται για μια σειρά από προβλήματα, πρόκειται για ε, τον πόλεμο στο Μαλί, πρόκειται για αλλαγές στο κλίμα και πρόκειται για ε, προβλήματα τα οποία ξεκίνησαν το 2012, είχαμε την επανάσταση των Τουαρέκ, είχαμε το πραξιβότημα στο Μαλί, έχουμε την ε, εντυνόμενη δράση του Μπόκο Χαράμ στην Νιγηρία ε, και έχουμε επομένως αυτή τη διατροφική κρίση στο Σαχέλ και επομένως ε, βλέπουμε πόσο ισχύει το ότι κανένα σχέδιο, κανένα πρόγραμμα, καμία θεωρία δεν μπορεί να, να ισχύει όταν είναι άσκηση επιχάρτου και βλέπουμε ότι τον Μάρτιο του 2011 επίσης είχαμε ε, τη στρατηγική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Είναι για ε, περιοχή μεγάλης γεωστατικής σημασίας έχει να κάνει με το, ενεργειακό μας πρόβλημα γίνεται επίσης εκεί πέρα διακίνηση παράνομη λαθρεμπόριο λαθρομετανάστευση περνάει από εκεί έχουμε επίσης εκεί και ο καταπολέμησης της τρομοκρατίας που πρέπει να μας απασχολήσει και ε, οπότε τώρα πρέπει να υπάρξει μια μακρόμνη στρατηγική ε, που να αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα, αγαπητοί συνάδελφοι, στα, στα καλύτερα σενάρια η στρατηγική της Ένωσης για το Σαχέλ θα πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση ε, τι μπορεί να κάνει με την παρέμβαση Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς πρόκειται να να χάσουμε κάθε έλεγχο, να χάσουμε κάθε αξιοπιστία όσον αφορά την αναπτυξιακή μας πολιτική. Έχουμε εδώ, και τέλο πάντων θα τον έχουμε ελπίζω σε, πολύ λίγο, τον, θα τον περιμένουμε τον κύριο Γενικό Γραμματέα του ΕΣΕΑΕ, τον κύριο Ποπόσκι. Θα συζητήσουμε μαζί του όλα αυτά τα καυτά ζητήματα. Να περιμένουμε ένα πεντάλεπτο προτείνω. Οπότε μπορούμε να ξεμουδιάσουμε να γίνει τελείως κατά αυτό το πεντάλεπτο Voilà, donc, euh, comme je vous le disais... Όπως έλεγα, έχουμε εδώ τον Γενικό Γραμματείο του ΕΣΕ, τον κύριο Ποπόφσκι, της ΕΕΛ στα ελληνικά. Να συζητήσουμε αυτά τα θέματα της καυτής επικαιρότητα. Σας ευχαριστούμε αγαπητέ κύριε που απεδέχτετε την ε, πρότασή μας. Σας δίνουμε για 15 με 20 λεπτά το λόγο. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για αυτή σας την ε, πρωτοβουλία, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας γιατί τώρα έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε γενικότερα τα ζητήματα για το Μαλί και για το Σαχέλ, να, να δούμε, να έχουμε γενική έποψη επομένω του τι γίνεται εκεί, πώ έχει εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για το Μαλί, μέσα στο Μαλί και όλα αυτά στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγής μας για το Σαχέλ. Και βεβαίω παρουσιάζει ενδιαφέρον για σας φαντάζομαι να δούμε πώς συνδέεται αυτού του είδου η συνολική προσέγγιση για το Μαλί και το Σαχέλ με τα όσα κάνουμε ε, σαν αναπτυξιακή πολιτική. Έχουμε εδώ τον ε, ε, συντονιστή μας για τα θέματα αυτά που υπηρετεί και εκείνος το ΕΕΔ και πήγε εκεί επί Οπότε μπορεί να σας πει περισσότερο για το πώς έχει η κατάσταση και τι προγραμματίζουμε να κάνουμε. Πρώτα πρώτα για το μαλλί, Η κατάσταση εξελίσσεται, είναι δυναμικού χαρακτήρα. Αλλάζει συνέχεια και όχι πλευρασμός μόνο ασφαλείας που είναι το, το πιο προβλημένο στην επικαιρότητα θέμα λόγω της παρουσίας της Γαλλίας, αλλά τελικά υπάρχει ένας χάρτης πορείας για, την, για ε, τον σχηματισμό της χώρας, εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, ε, είναι κάτι που μας αφορά όλους και θα πρέπει να ασχοληθούμε. Πρόκειται για ε, θέμα που συζητήθηκε στο Δουβλίνο από τους αρμόδιους υπουργούς. Συζητήθηκε από πολλές πλευρές, αλλά πάντως στα πλαίσια μιας τέτοιας σφαιρικής προσέγγισης και εμπλοκής, αυτό το οποίο θεωρήθηκε από τους υπουργούς ανάπτυξης τουλάχιστον το πιο σημαντικό ήταν το πώς θα μπορέσει να συνεχιστεί προς την περιοχή αυτή αυτή η αναπτυξιακή βοήθεια. Έχουμε αρχίσει να εκταμιεύουμε 250 εκατομμύρια ευρώ και δημοσιονομική υποστήριξη, βέβαια υπό όρους και προϋποθέσεις, θα σας τα πει εδώ και ο συνάδελφος, αλλά αυτό ε, ξεκίνησε από πολλές χώρες που είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι όροι και προϋποθέσεις, ας πούμε, το να δούμε πώς θα διεξαχθούν οι επικείμενε εκλογέ. Και τότε να χαμηλήσουν τα χρήματα πάντω, θα πρέπει να αποκατασταθεί η κρατική εξουσία σε βορρά και νότο. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι ε, το, αυτό που μας απασχολεί και ο Επίτροπος Πίμπαλξ συνεχίζεται σε επαφέ του ε, και σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ανάπτυξη αλλά βέβαια και οι Υπουργοί Εθνική Άμυνα ε, εδώ πέρα εμπλέκονται. Είχαμε βέβαια την ε, αποστολή μας στο Μάλι και την ανάπτυξη ε, των, των απεσταλμένων μας. Έχουν πάει εκεί 70 άνθρωποι μας, αυτοί που θα που τα μέσα Μαρτίου θα ξεκινήσουν την εκεί εκπαίδευση και κατάρτιση. Έχουμε αυτόν τον χάρτη πορεία επομένω. συνεργαζόμαστε με την Αφρικανική Ένωση, την ΕΚΟ, τα Ηνωμένα Έθνη, οπότε και συνεχίζουμε την εμπλοκή μας ε, για τα θέματα ασφάλεια. Έχουμε το UTM, έχουμε επίσης ε, την αφίσμα που είναι υποστήριξη προς ε, διάφορους ε, από διάφορε αφρικανικέ χώρε έχουν ήδη εκεί 4.000 άτομα στο Μαλί και στι γυρνιώσει χώρε. Το Ιε, ήδη εξετάζει το πώ θα ε, ε, γίνει αυτή η αποστολή να γίνει επιχείρηση του ΟΗΕ. Αυτό συζητείται, θα συζητηθεί στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω ακριβώ πότε, δεν γνωρίζω, όμως είμαστε σε επαφή με τον ΟΗΕ και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να ε, υποστηρίξουμε τον, τον στην προσπάθειά του. Υπάρχει εδώ και κάποιο άλλο στοιχείο ε, που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα, την τήρησή τους στο Μαλί. Συζητήθηκε το ζήτημα και από τα δύο συμβούλια και ανάπτυξης και υπουργού εξωτερικών και υπουργού ε, άμυνας και χθες κιόλα, γιατί έχουμε πλήρη επίγνωση του ότι εκεί έχουμε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους ε, στρατιώτες της χώρας ούτως ώστε να δούμε πώς θα υποπτεύσουμε την κατάσταση και να μπορέσουμε να έχουμε εκεί ανάπτυξη Αφρικανών και ανεξαρτήτων επίσης ε, παρατηρητών από μη οργανισμούς, οπότε ε, και ξεβρέθηκαν οι σχετικοί πόροι. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να αρχίσουμε ένα πρόγραμμα ανάκτησης ε, ούτω ώστε να έχουμε την ειρήνευση της χώρας, τη συμφιλίωση, την διαμεσολάβηση μεταξύ των διαφόρων ε, πλευρών στη χώρα και συγκεκριμένα στον, στο βόρειο τμήμα αυτή. Αυτή η κοινή αποστολή που σας ανέφερα πήγε στον Παμακό και εκεί διερευνήθηκε το τι χρειάζεται να γίνει, τι χρειάζονται οι αρχές, ε, να διαπιστωθεί τι θα πρέπει να γίνει, ποια σειρά, τι είδους μέσα πολιτικής θα πρέπει να μετέλθουμε και κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει κοινό προγραμματισμό. Το Μαλί, ξέρετε, το Μαλί ήταν ένα από του ε, υποψηφίου για κοινό προγραμματισμό και λόγω των πολιτικών εξελίξεων φρενάνε τη διαδικασία. Όμω ακόμα δεν έχουμε υπόψη τη χώρα γιατί θα πρέπει σύντομα να ξεκινήσουμε αυτό το κοινό πρόγραμμα για τη χώρα ε, σε συνεργασία με τα κρατη και προσπαθούμε τώρα να δούμε πώς έχει το όλο τοπίο. Προσπαθούμε να έχουμε μια συνολική, σφαιρική προσέγγιση, γιατί προσπαθούμε να δούμε ε, ε, τι, τι, τι θα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα ε, μετά, μετά τον, τον πόλεμο, με τι θα γίνει στο κέντρο της Αφρικής. Έχουμε ασχοληθεί με την περιοχή αυτή και προηγουμένως, όπως ξέρετε. Οπότε κατά κάποιο τρόπο τα θέματα είναι αλληλένδετα και έχουν σχέση και με την δέσμευσή μας να έχουμε μια συνεπή, συνεκτική πολιτική για την ανάπτυξη, γιατί ακριβώς εκεί ε, συνδυάζουμε ε, διάφορα μέσα πολιτικής, πολιτική εμπλοκή, ε, μακροπρόθεσμα μέσα, πρόθεσμα την, την, την, την, δέσμευση της, μας για τις προσπάθειες και πάρα στα πλαίσια του Ταμείου Ανάπτυξης και στον Νίγηρα επίσης έχουμε κάνει εκπαίδευση ε, χωροφυλακής, αστυνομίας ε, για την περιοχή. Και αυτό που με ενδιαφέρει να ακούσω τις δικές σας σκέψεις. Πώς εσείς σχετίζετε όλα αυτά την υλοποίηση της στρατηγικής μας για, για το Σαχέλ ε, με την ανεπτυξιακή μας πολιτική. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, μπορεί να σας πει εδώ ο συνάδελφος να σας μιλήσει για την αποστολή του στο Μαλί. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον. Uh, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ Μάτσι. ήθελα και εγώ να σας πω ορισμένα πράγματα σε σχέση με την έκβαση της υπηρεσιακής ε, αποστολής στην Παμακό ε, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της έγκρισης του οδικού χάρτη από την Εθνική Συνέλευση του ε, Μαλή. Όταν φτάσαμε εκεί, τη στιγμή της ενδεχόμενης έγκρισης στην Παμακό, θέλαμε να δείξουμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πολιτική παρουσία και πολιτική δέσμευση ε, με το Μαλί σε σχέση με το πολύ σημαντικό αυτό θέμα, το οποίο, ε, σημαντικό βήμα το οποίο έπρεπε να κάνει η Εθνοσυνέλευση. υπηρεσιακή αποστολή σημαίνει ότι η σύνθεση ήταν από την ΕΡΙΕΔ, διάφορα τμήματα της ΕΡΙΕΔ, ε, από τα γεωγραφικά γραφεία και τη γεωγραφική παρουσία ε, και από το ε, Τμήμα Πολιτικής για τη Διαχείριση των Κρίσεων, το CMPD, συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ, όπως επίσης και εκπροσώπηση από τα κράτη-μέλη. Βασικά η σύνθεση ήταν πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια περιεκτική προσέγγιση, τι πρέπει να γίνει σε ε, βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα για να υποστηριχθεί ο χάρτης πορείας ε, όπως εγκρίθηκε, όπως αυτό εγκρίθηκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να ε, κινηθεί σε τρεις ε, παράλληλες οδούς, συμπέρασμα, σύσταση της διυπηρεσιακής αποστολής στην Μπαμακό, βραχυπρόθεσμα, μακρυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Έχουμε και τρία διαφορετικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτές τις πορείες. Κάθε ένα από αυτά έχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την λήψη των αποφάσεων, για την εφαρμογή τους και ε, βέβαια μια διαφορετική ε, προοπτική ε, προετοιμασίας. Πρώτα υπάρχει το μέσο σταθερότητας, ε, γιατί είναι ε, ένα από τα πρώτα που μπορούν να επιφέρουν αποτελέσματα. Το τι αποτέλεσμα θα θέλαμε να έχουμε μέσω του μέσου σταθερότητας ε, στο Μαλί, το πρώτο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι η υποστήριξη της ε, πολιτικής διαδικασίας συμφιλίωσης, άμεση υποστήριξη στην εφαρμογή του χάρτη πορείας, βράχη πρόθεσμα, ε, έναρξη προετοιμασίας για τις εκλογές, όπως επίσης ε, και υποστήριξη στις ανακτημένες περιοχές, περιοχές που ανακτήθηκαν από τη στρατιωτική παρουσία και από, τους διάφορες, από την παρουσία διαφόρων στρατιωτικών ομάδων, κυρίως στο Βορρά. Αυτό που θέλουμε λοιπόν να δούμε ε, μέσω, του, ε, μέσω σταθερότητας είναι ε, να έχουμε μια κοινή προσέγγιση στο βορρά και στο νότο και αυτό είναι ένας γνώμονας ε, στη δέσμευσή μας ε, με το Μαλή, όχι μόνο για το μέσο σταθερότητας αλλά και για άλλα μέσα που θα τα αναφέρω ε, εντάχει. Αυτή η παράλληλη προσέγγιση πρέπει να είναι ένας γνώμονας, μία αρχή που θα μας καθοδηγεί. Τώρα, η επανέναρξη της αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτό έχει να κάνει με το ε, Ταμείο Ανάπτυξης γιατί λόγω της στρατιωτικής επίθεσης και λόγω των προβλημάτων που υπήρξαν των δυσκολιών στο, στο Βορρά σταμάτησε αυτό το πρόγραμμα και πρέπει να ε, αναβιώσει ώστε να μπορέσουμε να ε, υποστηρίξουμε την επιστημιστική ασφάλεια, την υδροδότηση, την εκπαίδευση, ε, τα κοινωνικά προγράμματα, όχι μόνο στο Νότο, αλλά και στο Βορρά. Αυτό είναι το δεύτερο, η δεύτερη μας ε, οδός, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε εκ νέου αυτά που είχαν ήδη δρομολογηθεί, όμως με μεγαλύτερη έμφαση στο βορρά από ό,τι στο παρελθόν. Τρίτο στοιχείο είναι κατά τη πιο μακροπρόθεσμο, αλλά πρέπει να ορίσουμε και τι θα πει μακροπρόθεσμο για το μαλλί. Μέχρι το τέλος ε, της χρονιάς ε, υπάρχει μία πρόταση της διπηρεσιακής αποστολής να υπάρχει ε, ένα συμβόλαιο οικοδόμησης κρατικής υποδομής, ώστε να δείξουμε ότι μπορούμε να απαντήσουμε ε, σε μια χώρα, να ανταποκριθούμε σε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίση. Ε, αυτή η ιδέα θα δοκιμαστεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε πώς μπορούν ε, να υποστηριχθούν οι προσπάθειες με τη χρήση αυτού του μέσου. Κάτι τέτοιο βέβαια μπορεί να χρειαστεί κάποιο χρόνο προκειμένου να συζητηθεί, να αναπτυχθεί και να επιτύχει την ουσία των στόχων. Ε, νομίζω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε καλύτερα να, να εξηγήσει τι είδους χρονοδιάγραμμα μπορούμε να ε, προβλέψουμε όμως δεν θα πρέπει να είναι μια παρατεταμένη διαδικασία ή μια διαδικασία που θα αναβληθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ίσως θα έπρεπε ένα χρονοδιάγραμμα ε, να εγκρίνουμε το οποίο θα ε, λέει ότι στους πρώτους έξι μήνες του, του έτους του 2013 πρέπει να επιτευχθούν τα αποτελέσματα αυτά για την οικοδόμηση των κρατικών υποδομών. Επίσης συζητήθηκε και αναφέρεται και στο, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ότι θα υπάρξει και μία έκκληση διάσκεψης δωρητών ε, το, την Άνοιξη, κάτι το οποίο είναι ένα επιπλέον στοιχείο που θα ε, αποτελεί τμήμα ε, της περιεκτικής μας προσέγγισης στις δραστηριότητές μας στο Μαλί αξιολογήσαμε εμείς ε, τις ανάγκες ε, της κυβέρνησης ε, των πολιτών και των πολιτικών συγκυριών του Μαλή στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χάρτη πορείας και τα παρουσιάσαμε στις υπηρεσίες μας, τις βασικές αρχές τουλάχιστον και το κύριο περιεχόμενο της πρότασης αυτής. Νομίζω ότι το μέσο σταθερότητας ήδη ε, έδρασε και λήφθησαν αποφάσεις την περασμένη εβδομάδα, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι η δυναμική αυτή βοήθησε να υπάρξει η πρώτη δράση επιτόπου χθες, όπως είπε και ο Μάτσεϊ, η ιδέα αυτού του συμβολέου οικοδόμησης κρατικών υποδομών συζητήθηκε και με τους Υπουργούς Εξωτερικών Υποθέσεων και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο ώστε να αναπτυχθεί κατά τέτοιο κατά τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κιόρενς ως μόνιμος εισηγητής για τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Ποπόφσκι και τον εμπειρογνώμονά του για τα θέματα που αφορούν το Μάλι. Σας ευχαριστώ για την ε, έκθεσή σας σχετικά με την ολιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση στο Σαχέλ και πιο συγκεκριμένα στο Μάλι. Κάποιες ερωτήσεις αρχικά. Και μετά θα κάνω και σχόλια. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων συζητήθηκαν θέματα όπως Σεουδική Αραβία και Κατάρ που, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι υποστηρίζουν τα τρομοκρατικά δίκτυα στις ε, περιοχές αυτές. Και αν ναι, τι αντιδράσεις ε, παρατηρήθηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων. Δεύτερον, για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις υποθέτω και δεν είμαι ο μόνος φαντάζομαι που έχω τέτοιου είδους προβλήματα ότι αυτή η δράση εντάσσεται στα πλαίσια του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Τα Ηνωμένα Έθνη πριν από την γαλλική παρέμβαση είχαν αποδεχθεί την αρχή μιας στρατιωτικής παρέμβασης δυνάμεων της ε, CDAO, της, ε, των δυνάμεων της, Ανατολικής, ε, της Δυτικής συγγνώμη, Αφρικής. Και επειδή πίεζε ο χρόνος, το Μάλι ζήτησε από τη Γαλλία να παρέμβει. Δηλαδή, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αυτή η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Επόμενο ερώτημα. Για τα θέματα διεθνούς δικαίου, τα δύο κράτη-μέλη που έχουν δικαίωμα βέτος στο Συμβούλιο Ασφαλείας εξηγούν τη θέση τους στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ή όπως στο παρελθόν δεν συζητούνται τέτοια θέματα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Έγινε κάποια ανταλλαγή απόψεων και ποιες ήταν οι αντιδράσεις των κρατών μελών. Αυτές είναι οι πρώτες μου τρεις ερωτήσεις και έχω και μια τέταρτη στη στρατιωτική δράση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλοί διαπίστωσαν ότι η Γαλλία μάλλον μόνη της φάνηκε να είναι. Ε, μας λένε ότι το Μάλι ζήτησε από τη Γαλλία να παρέμβει. Το Μάλι έκανε μια έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση, πιστεύω. Κατά τα άλλα, άκουσα πολύ προσεκτικά με μεγάλο ενδιαφέρον τη στάση τη Ευρωπαϊκής Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε αυτή τη φάση της κρίσης. Και νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε για τις ενδεχόμενες δυνατότητες που υπάρχουν και κάποια όρια τα οποία δεν πρέπει να ξεπεράσουμε ή τέλος πάντων κάποια σημεία πέρα από τα οποία δεν πρέπει να φτάσουμε. η δράση της κυρίας Γεωργίευα πιστεύω ότι ήταν πραγματικά υποδειγματική. Παρενέβη υποδειγματικά και χθες την παρουσία της εδώ πολύ το τονίσαμε. Νομίζω ότι η κυρία Γεωργίευα παρενέβη με θάρρος διότι υπερασπίζεται στεναρά και εμείς την υποστηρίζουμε την αρχή της αμεροληψίας. Πράγμα το οποίο, όπως είπατε, δεν εμποδίζει το να δημιουργηθούν, το να λάβουν χώρα ε, συνεδριάσεις μεταξύ υπηρεσιών στον Παμάκο. Δηλαδή μπορούμε να συνδυάσουμε την αμεροληψία με την βούληση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και αυτό επιβεβαιώνει την ε, απόλυτη τήρηση της αρχής της, αμεροληψία. της ε, αμεροληψίας. Σωστά λέτε ότι πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου. Η πιο σημαντική δουλειά και με τα πιο μόνιμα αποτελέσματα γίνεται στον τομέα που είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, την διοίκηση Κοντεφ, για τις εκεί δράσεις και εδώ θα πρέπει να τηρήσουμε την αρχή της εταιρικής σχέσης. Θα ήθελα όμως να μου πείτε γιατί δεν θέσαμε περισσότερο έντονα το θέμα της έλλειψης ασφάλειας στο Μάλι. Ε, και ως Υπουργός ε, Αναπτυξιακής Συνεργασίας είχα προγράμματα στο Κιντάλ και θυμάμαι τότε το 2002 μου είχαν πει να μην πάω σε αυτή την περιοχή διότι αυτό ήταν διπλωματικό πεδίο και η πρεσβεία ε, των κάτω χωρών που εκπροσωπούσε τότε και εκπροσωπεί και τώρα τη χώρα μου στο Μάλι μου είχε πει να μην πάω εκεί για επίσημη επίσκεψη για λόγους ασφαλείας. Ξέρουμε πόσο δύσκολο ήταν να γίνουν διακανονισμοί μεταξύ των δυνάμεων των επαναστατών και της κεντρικής εξουσίας στον Παμάκο και νομίζω ότι τελικά μπορούμε να πούμε ότι κάπως ξεπεράσαμε τις δυσκολίες θέτοντας πρώτων ευθυνών τους τους του ΑΡΕΓ και ζητώντας τους να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και στην κυβέρνηση. Τι συνέβη στη χώρα αυτή στην οποία ήμασταν έτοιμοι ε, να προγραμματίσουμε το μέλλον, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, τι έγινε ε, που οδήγησε αυτή η χώρα στη ρήξη. Η στρατηγική την οποία ακολουθήσατε το 2011, το Μάρτιο αν θυμάμαι καλά, ήταν επαρκής για την πρόληψη αυτής της κρίσης. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι που μας έφεραν προς προτετελεσμένου γεγονότος. Αυτές τις παρατηρήσεις είχα. Αφήνω το λόγο στους συναδέλφους και στο τέλος ελπίζω να μου ξαναδώσετε το λόγο για να κλείσω. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον κύριο Μπέρμαν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο κύριος Μπέρμαν, για αυτά τα οποία τόσο ξεκάθαρα μας εξηγήσατε για το τι κάνετε και τι προγραμματίζετε να κάνετε και θα περιοριστώ προσωπικά σε ένα σημείο χρειάζεται να ξανααποκτήσει η χώρα το Μαλί αποδεκτή διακυβέρνηση. Λέει, λατήθηκε η χώρα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να διοικηθεί τώρα. χρειάζονται επενδύσεις. Μας είπατε κύριε Ποβόσκη για δημοσιονομική στήριξη πάρα πολλέ ε, χώρες, αλλά και η δική μου χώρα, η Ολλανδία, διστάζουν πάρα πολύ να προβούν σε τέτοια κίνηση. Γι' αυτό και δεν είναι πλάκι. Πάντως. Εάν θέλουμε διοίκηση, κυβέρνηση που να λειτουργήσει χρειάζεται και χρήμα. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με τη δημοσιονομική στήριξη, αλλά θα ήθελα να μου πείτε συγκεκριμένα ποιε είναι οι προϋποθέσεις, ποιοι είναι οι όροι που έχετε τάξει για να χορηγηθεί αυτή η βοήθεια. Επίσης θα ήθελα να μάθω κατά πόσον διατίθεται κάποιο ποσόν προκαθορισμένο που να θεωρείται το, το, το, το, όργανο, το μέσο πολιτικής για αυτή τη στήριξη. Ευχαριστούμε κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ποπόφσκι. Όντως, πριν από δύο μέρες ε, ε, είχαμε την ευκαιρία να δούμε την κυρία Γεωργίευα, τον, τον ε, Πρωθυπουργό της χώρας, οπότε και το θέμα φωτίζεται τώρα διαφορετικά από εσά. Γιατί αυτές οι τρεις συναντήσεις ήταν πάρα πάρα πολύ ωφέλιμες. Πρώτα πρώτα. Πρόληψη και παρέμβαση-επέμβαση. Πρόσφατα αυτούς τους τελευταίους μήνες η υπηρεσία εξωτερικής δράσης έχει ορθά ενεργήσει όσον αφορά την διαχείριση των κρίσεων, αν μπορούμε αυτό να το πούμε, ε, να χρησιμοποιηθεί την έννοια ε, στην ευρύτερη της ε, σημασία. Δόθηκαν οι δέουσες απαντήσεις στην κρίση. Και σήμερα αυτό το οποίο έχουμε αποδεικνύει την ορθότητα των ενεργειών. Ο Σάρλ είπε κάτι προηγουμένω το οποίο έχει να κάνει με την ε, πρόληψη και ακριβώ έχουμε ε, το θέμα του πώς η πολιτική μας θα καλύψει και την πρόληψη. Ναι, μπορούμε να πάμε για την ασυγκρότηση της χώρας κλπ. λοιπά Και υποθέτουμε ότι όλοι θα βοηθήσουν και ενδιαφέρονται. Όμως υπάρχει ένα άλλο σενάριο. να έχουμε ανταρτό πόλεμο. Να έχουμε τρομοκρατία που να χτυπήσει ξανά και ξανά και επανειλημμένα. Και ας πούμε ότι το Μάρτι ή ξέρω εγώ πότε, όποτε προβλέπετε να φύγουν οι εμπλές γαλλικές δυνάμεις. Τι θα γίνει με την κατάρτιση, την εκπαίδευση. Πώς εκπαιδεύεται εκεί πέρα τις ένοπλες δυνάμεις, για παραδοσιακό πόλεμο ή για αυτό το οποίο... Γιατί ακριβώς πρόκειται για τελείως διαφορετικούς πολέμους που συμβαίνουν. Πρέπει κάτι να γίνει επομένως από πλευράς πρόληψης. Να σκεφτούμε και αυτό το σενάριο, το οποίο δεν είναι καθόλου απίθανο κάτι άλλο τώρα που θέλω να επανέλθουμε είναι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συγκεκριμένα των ανηλίκων, των, των γυναικών για αυτές τις, την τραγωδία που, που έχει συμβεί στη χώρα. Εκεί είναι καθημερινό φαινόμενο. Η πάση ε, οι βιασμοί και δεν είναι μόνο οι επαναστάτες, μόνο οι, οι, οι αντάρτες. Όλοι, όλοι εγκληματούν κατά αυτόν τον τρόπο. Με ατιμορρησία. Είδαμε τι έγινε στο Κονγκό. Όλοι είχαν ευθύνε. Μας μιλήσατε για μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έγινε αυτή η συνάντηση με το βουλευτή που έρχεται σε επαφή με τις μη οργανώσεις που ασχολείται, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτού του είδους η ατιμωρησία θα πρέπει κάποιος να φροντίσει αυτές τις, τα θύματα τόσο, της γυναίκας, τα θύματα των βιασμών, ε, γιατί μιλάμε για τη δέσμευσή μας. Τη δέσμευσή μας να ανασυγκροτήσουμε τη χώρα. Και σε αυτά τα πλαίσια δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η ατιμορρησία. Ναι, μιλάμε για δικαστήρια, για δίκες. Δεν νομίζω ότι είμαι η μόνη που θέλει να υπάρξει έλεγχος γιατί αλλού που είχαμε τέτοια φαινόμενα αποτύχαμε παταγωδός. Και κάτι άλλο κύριε Ποπόφσκι. Στην τρέχουσα συγκυρία όλοι λέμε για το τι θα γίνει ο πλευρά ε, υπηρεσία εξωτερική δράση και μα είπατε για αυτέ τι κοινέ υπηρεσίε κλπ. κλπ. Μήπω μπορείτε να μου πείτε στα πλαίσια τη λειτουργία τη υπηρεσία αυτή ποιε είναι. Τι γίνεται, πώς λειτουργεί αυτό το σχήμα που είπατε. Να έχουμε διαφάνεια. Ε, είναι μόνο η διεύθυνση που, που, κάνει, που είναι αρμόδια για την διαχείριση των κρίσεων. Ε, τι ακριβώς γίνεται, πώς, πώς, πώς λειτουργεί το, η υπηρεσία σε αυτό το μέτωπο. Ευχαριστούμε. Κύριος Νάιζερ τώρα ζητεί το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Ε, νομίζω ότι είναι εσφαλμένη η στάση μας έναντι της διαδικασίας εκδημοκρατισμού του Μάλι και πρέπει να αναρωτηθούμε πώς φτάσαμε σε αυτή τη λάθος εκτίμηση. Ο συνάδελφος Γκέρενς επίσης το ανέφερε ε, γιατί ήταν γνωστό ότι υπήρχε αστάθεια στην ε, χώρα και όταν μιλάμε για μια περιφερειοποίηση στο Μάλι, οι προσπάθειε ήταν πάρα πολύ αόριστε. Πριν από δύο χρόνια είχα πάει στον Παμάκο και ο στόχο ήταν η κοινωνία των πολιτών, οι τοπικές αρχές, οι αρχές αυτοδιοίκηση, η αποκέντρωση, κάποια προγράμματα τα οποία ε, δεν είχαν ε, ακόμη επίπτωση, δεν είχαν ε, πραγματικά αποτελέσματα επιτόπου και μετά την σύραξη στη Λιβύη ήταν πολύ εύκολο να φανταστεί κανείς πώς θα μπορούσε ε, ε, να κλιμακωθεί η κατάσταση και στο Μάλι και για το ECOVAX υπάρχουν πολλές κριτικές διότι ε, θεωρήθηκαν δύναμη εισβολής από τους ε, πολίτες στο Βορρά. Και πρέπει να δούμε ποια ήταν τα μέσα άμεσης ανάγκης που θα έπρεπε να λυθούν για να υπάρξει η δυνατότητα αποδοχής τους από τους του ΑΡΕΓ. Νομίζω ότι ε, ε, θα πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε τις διαφορές που υπάρχουν ε, και μεταξύ κυβερνήσεων και μεταξύ στρατιωτικών δυνάμεων ε, όσον αφορά τους Ευρωπαίους, διότι υπάρχουν διαφορές και είναι πολλή η δουλειά που πρέπει να γίνει και από πλευράς Ευρωπαίων. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συντομότερο δυνατόν να φτάσουμε σε νέες εκλογές στο Μάλι. Ευχαριστώ πολύ θα λάβω για λίγο το λόγο για να υποστηρίξω αυτά που είπε και η κυρία Ντεκάιζερ κατά των εγκλημάτων, κατά των βιασμών που είναι ζητήματα που μας απασχολούν είτε πρόκειται για περιοχές σύραξης είτε όχι. Μπορεί να τα καταγγέλουμε όλα αυτά οπουδήποτε και αν συμβαίνουν αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να χτυπήσουμε το χέρι μας στο τραπέζι και να πούμε ότι δεν ανεχόμεθα τέτοια εγκλήματα. Συνήθως δείχνουμε μεγάλη επίοικια προς τα εγκλήματα αυτά. Είναι καταστροφικά όχι μόνο για γυναίκες, μιλάμε και για μικρά κοριτσάκια εγώ πιστεύω ότι δεν είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί, ίσως διότι δεν είμαστε αρκετά απαιτητικοί. Ευχαριστώ. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ποπόφσκι και μετά στον κύριο Γκέρενς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύνθετο το θέμα. Θα προσπαθήσω να, να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις ε, και όλα τα σχόλια. Ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ δεν συζητήθηκε από τους Υπουργούς. Παρακολουθούμε ε, την κατάσταση, παρακολουθούμε τα γεγονότα, αλλά δεν ε, έγινε ιδιαίτερη συζήτηση από αυτού. Όντως υπάρχει μια στρατιωτική παρέμβαση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, και είναι το ψήφισμα 2085 του Συμβουλίου Ασφαλείας το σημείο στο οποίο ε, στηριζόμαστε και για τη γαλλική ε, επέμβαση και για την επέμβαση της αφίσμα της ε, Αφρικανικής Αποστολής. Η Γαλλία ήταν σε επαφή μαζί μας στην φάση προγραμματισμού, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μας εξέπληξε η γαλλική παρέμβαση, είναι μια γαλλική προσπάθεια, αλλά υπήρξε υποστήριξη για την επέμβαση της Γαλλίας και πρακτική υποστήριξη από τα κράτη-μέλη μονομερός, την οποία εμείς παρακολουθήσαμε όσο προχωρούσε αυτή η κατάσταση και μέσα στο στρατιωτικό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε παρακολούθηση. Η κυβέρνηση του Μάλι απευθύνθηκε στη Γαλλία, ζήτησε βοήθεια από τη Γαλλία. Αυτό ήταν ο άμεσος λόγος για την παρέμβαση της Γαλλίας. Είχαμε ανταλλαγέ απόψεων με το ΕΚΟΒΑΣ και με το Μάλι για ε, υποστήριξη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους εκπαίδευση. Δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων ε, επιταχύναμε αυτή την αποστολή εκπαίδευσης και ελήφθη χθε η απόφαση να ξεκινήσει αυτή η αποστολή παρότι μας έλειπαν ακόμη κάποια σημεία όσον αφορά τις δυνατότητες που έχουμε. Τελευταία στιγμή, ακόμη και χτες, αναζητούσαμε ελικόπτερα για ε, η ιατρική διακομιδή. πάντω τα καταφέραμε ακόμη και τελευταία στιγμή να το οργανώσουμε. Συμφωνώ κύριε Γκέρεν, για αυτό το οποίο είπατε για τη δράση τη Επιτρόπου Γεωργίευα. Ήταν πραγματικά υποδειγματική και όντω ενεργεί με βάση τις αρχές της ανθρωπιστικής παρέμβασης. Αυτές είναι οι αρχές της αμεροληψίας και της ουδετερότητας που πάντοτε τηρούμε. Ό,τι και να κάνουμε γνωρίζουμε ότι ο ανθρωπιστικός άξονας, οι ανθρωπιστικές δράσεις χρειάζονται χώρο. Εμείς τα συντονίζουμε και ξέρουμε ότι πρέπει να δίδεται πρόσβαση και πρέπει όλοι να τηρούν την αρχή της ουδετερότητας, πράγμα το οποίο κάνουμε και εμείς. Για τη στατική για το Σαχέλ θα ζητήσω από τον Πέτερ να σχολιάσει και για τα θέματα πρόληψης. Προς τον κύριο Μπέρμαν, βεβαίως και θα επικεντρωθούμε στην αποκατάσταση της διακυβέρνησης και δεν είναι κάτι καινούριο ότι ορισμένα κράτη-μέλη είναι λίγο περισσότερο διστακτικά όταν μιλάμε για δημοσιονομική υποστήριξη και ο Ολλανδός Υπουργός το Δουβλίνο το είπε. Πάντως ε, όλοι συμφώνησαν ότι θέλουμε να βοηθήσουμε την αποκατάσταση της ειρήνης και υπάρχουν κάποιοι όροι. Κάποιες ε, χώρες έκαναν σαφή σύνδεση με το θέμα των εκλογών. Οι εκλογές ε, ε, υποτίθεται ότι θα γίνουν τον Ιούλιο και ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθούν οι εκλογές μπορεί επίσης να είναι καθοριστικός για την εκταμίευση ποσών και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί. Ο κύριος Νόιζερ επίσης μίλησε για τις εκλογές. Θα υποστηρίξουμε την προετοιμασία των εκλογών και θα στείλουμε και μία αποστολή παρατήρησης των εκλογών στο Μάλι με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως κάνουμε συνήθως. Ήδη από τώρα θα αρχίσουμε λοιπόν να κάνουμε τον προγραμματισμό, γιατί δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Τώρα για την απειλή ανταρτοπολέμου που ανέφερε η κυρία Ντεκάιζερ, όντως είναι μια υπαρκτή απειλή και δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας με την αποστολή μας για την εκπαίδευση του στρατού. Θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τις εγχώριες δομές για την επιβολή του νόμου, την αστυνομία, για το στρατό κλπ και την περασμένη εβδομάδα το συζητήσαμε ένα ποσό 20 εκατομμυρίων που διατίθεται ως βοήθεια θα πάει στην υποστήριξη αυτών των φορέων. Εξοπλισμός, οχήματα για να μπορούν να λειτουργήσουν. Παράλληλα όμως αυτό το οποίο προβλέπουμε και έχει αρχίσει η διαδικασία προγραμματισμού γι' αυτό είναι το να επεκτείνουμε ενδεχομένως μία αποστολή εκπαίδευσης μη στρατιωτικού προσωπικού, κάτι που ξεκίνησε στον Ήγηρα και μπορεί να επεκταθεί και στο Μάλι. Δεν μπορώ να σας πω πότε θα γίνει, αλλά είναι τμήμα του μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου προγραμματισμού μας. Ήδη έχουμε έναν αξιωματικό σύνδεσμο που είναι τοποθετημένο στην αντιπροσωπεία μα στο Μπαμάκο, και θα αρχίσουμε τη διαδικασία προγραμματισμού. Και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε με τις υπηρεσίες ασφαλείας και δικαιοσύνης στο Μάλι. Όλοι αντιλαμβανόμαστε γενικότερα και το συζητήσαμε και με τον Επίτροπο Πίμπαλξ ότι η ασφάλεια είναι ένας σημαντικός τομέας παρέμβασης. Όλο και περισσότερο λοιπόν εξετάζουμε την ασφάλεια και για τις χώρες του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας και για τις χώρες ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Δεν μιλάμε για εξοπλισμό του στρατού, αλλά μιλάμε για επένδυση στην ανάπτυξη θεσμών. Όσον αφορά την ατιμορρησία, και αυτό είναι κάτι που θα αποτελέσει έναν από τους όρους που θα θέσουμε όταν συμφωνήσουμε με το Μάλι οι υπηρεσίε ήταν οι γεωγραφικέ υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τη Επιτροπή, ε, το τμήμα ε, αντιμετώπιση κρίσεων τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και ιδιαίτερα το τμήμα ασφάλεια και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με την μεσολάβηση, γιατί εξετάζουμε και τη δυνατότητα μεσολάβηση μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων στο Βορρά, των Αράβων και των Τουαρέγ. και το τμήμα των προγραμματιστών μας ε, από το τμήμα CPCC, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται. Όσον αφορά την προοπτική για αποστολή Ηνωμένων Εθνών, αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσουν τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά έχουμε τακτικά συζητήσεις μαζί τους. Έκανα εγώ μια συνάντηση με τον κύριο Λατσούχο, επικεφαλής ε, του Τμήματος ε, Διασφάλισης της Ειρήνης. Κάναμε μια συνάντηση στο Δουβλίνο την περασμένη εβδομάδα δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ελπίζουν ότι θα υπάρξει κάποιο νέο ψήφισμα ή κάποια δήλωση του Πρόεδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου ε, για να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαν να μπουν οι αφρικανικές δυνάμεις υπό τη σημαία του ΟΗΕ. Αυτό όμως μπορεί να απαιτήσει κάποιους μήνες. Ε, είμαστε έτοιμοι να το υποστηρίξουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη για να μας πούν τι περιμένουν από εμά για να τους βοηθήσουμε. Πρόεδρε, να ζητήσω από τον Πέτερη να παρεμβεί για τα άλλα σημεία που αναφέρθηκαν. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομο. Ε, πλέον σχόλια από πλευρά. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την ε, αποστολή μα, ε, θα πρέπει να σα τονίσω ότι πρόκειται για μια αυθεντικά εταιρική σχέση μεταξύ όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών στην εξωτερική υπηρεσία, εξωτερική δράση, Κομισιόν, ΕΚΟ, κράτη-μέλη ε, επομένως, πρόκειται για κάτι ε, οριζόντιου χαρακτήρα. Συμμετέσχουν όλοι, όλοι, όλοι σε αυτήν την αποστολή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο είδους ε, αξιολόγηση, γιατί θέλαμε μια τέτοια διακλαδική αποστολή, όχι μόνο για να βρούμε τους πιο καλούς τρόπους, τους πιο σωστούς τρόπους, να δούμε τι θα κάνουμε βράχη και μάκρο πρόθεσμα, αλλά επίσης να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο πώς θα έχουμε έναν κοινό προγραμματισμό και κάθε τον τρόπο προσπαθούμε να δούμε ε, πώς θα προλιάνουμε το έδαφος για όλα αυτά τα οποία προαναφέρθησαν σε σχέση με την αρχική ιδέα, το πώς δηλαδή το Μαλί θα είναι μία από τις χώρες ε, όπου μπορεί να έχουμε έναν κοινό προγραμματισμό και η, όλη αυτή η διαδικασία ε, είχε τους επικεφαλής των αντιπροσωπιών στο τιμόνι και πρόκειται επομένως ε, για κάτι τέτοιο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε ε, πώς θα έχουμε ανάληψη ευθυνών, δέσμευση σε σχέση με τις αρχές. Τώρα κάτι άλλο όσον αφορά ε, τη στατική μας για το Σαχέλ. Συζητώντας αυτό το ζήτημα και συζητώντας το με τις αρχές της χώρας, με τους εκπροσώπους της χώρας σε αυτή την περιοχή σε σχέση με ε, τους, τους εταίρους μας στην περιοχή. Καταλήφθω ότι έχουμε τρία-τρία στοιχεία σε σχέση με το πώς φτάσουμε στην κλιμάκωση. Έχουμε τον εξωτερικό παράγοντα, έχουμε ε, παρουσία εξωτερικού παράγοντα ε, και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ε, κάποιο είδου φαινόμενο χιονοστιβάδας σε σχέση με το πώς ξεκίνησαν όλα στην Λιβύα και τελικά σε πάρα, πολλές, πάρα σημεία της χώρας ε, και κυρίως στον Βορρά ε, έγινε μια τέτοια ε, ένταση του φαινομένου. Επίσης έχουμε και την, την παράνομη διακίνηση ανθρώπων και όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο οδηγούν σε, σε πραξικόπημα, οδηγούν σε στρατιωτική δράση στον Βορρά. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πάμε στο τι έγινε προ δεκαετίας. Άρα γι' αυτό θα πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, να μην κάνουμε τα ίδια λάθη εκείνα τα οποία ήδη ε, προηγήθηκαν, αυτά τα οποία ε, ήδη κάναμε. Τώρα, τη στρατηγική για το Σαχέλ, δεν ε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα έχουμε από το εξωτερικό φαινόμενο της χιονοστιβάδας όταν εγκριθεί η στρατηγική μας, αλλά πάντως υπάρχει κάποιο είδους διακυβέρνηση ε, η οποία είναι μάλλον αδυναμητρό όσον αφορά το, το συμβόλαιο, τη σύμβαση, τη δέσμευση για την συγκρότηση του κράτους. Όπως προείπα, πρόκειται για ένα τελείως ε, νέο μέσο πολιτικής, κάτι το οποίο τώρα προκύπτει από την ανακοίνωση η οποία εξεδόθη το 2011 για την δημοσιονομική στήριξη. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς έτσι θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες τους. Και θα πρέπει μενός κάπως να δούμε αυτή την πτυχή, τη, τη, συμβατική. Δεν είναι κάποιο είδους κλασική δημοσιονομική στήριξη. Πρόκειται να έχουμε εδώ και την πτυχή της ασφάλειας, κάτι το οποίο μας αφορά όλους ακριβώς, γιατί έχουν ε, μπει και κάποιες προϋποθέσεις και όρια σε αυτό το συμβόλαιο. Και θα πρέπει επίσης να δούμε τι είδους εξελίξεις έχουμε ε, να δούμε πώς είναι δυνατόν να έχουμε πληρωμή, βοήθεια, σε δόσεις και όχι εφάπαξη. Και έτσι, τέτοια, τέτοια προσέγγιση θέλουμε. Οπότε για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την παρακολούθηση και υποπτία των όσων γίνονται, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με όρου και προποθέσει, τι εξελίξει έχουμε επιτόπου και πού πάει το πράγμα. Πρόεδρο. Έχουμε πάρα πολύ καθυστερήσει. Έχουμε ακόμα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη. Ο κύριο Γκέρεν πρέπει να πάρει το λόγο για να συνοψίσει. Οπότε, κύριε Μπέρμαν, δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σα. Έχετε σχόλια για την επιβεβαίωση του Φρονσουά Ολόγκο ότι 7 πολίτες Γάλλοι ε, έπεσαν θύμα απαγωγή στο Βόρειο Καμερούν. Σήμερα το πρωί αυτό. Ναι, είναι γεγονός αυτό, το γνωρίζουμε αλλά γνωρίζουμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι τώρα είναι πιο εκτεθειμένοι σε απαγωγές και σε ομοιρία σε σχέση με το παρελθόν. Εντάξει, θα το προσθέσουμε στο χρονοδιάγραμμά μας, στον προγραμματισμό μας, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Γκέρεν τώρα για να συνοψίσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τέσσερα σημεία συμπερασματικά. Πρώτον, αυτό που κάνουμε δεν είναι αρκετά ορατό. Έχουμε πρόβλημα ορατότητα. Αυτό που φάνηκε στο Μαλί ήταν η γαλλική παρέμβαση. Αυτό που κάνουμε στα, στο ανθρωπιστικό τομέα και στον αναπτυξικό τομέα δεν είναι αρκετά, γνωστός, ε, αρκετά γνωστό. Δεν είναι το, το σημαντικότερο, αλλά τέλο πάντων είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δέχεται ο Ευρωπαίο φορολογούμενο ε, καλύτερα τι πολιτικέ μα και τι αποφάσει μα. Το Μαλί δεν είναι μόνο διεθνέ πρόβλημα, είναι και περιφερειακό πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναπτύξουμε περισσότερο την περιφερειακή διάσταση. Μιλήσατε για το εφέ το ντόμινο, του ντόμινο. Ε, και απαντήσατε και στην κυρία Ντεκάιζερ ε, τώρα στο Καμερούν το βλέπουμε να, να το το εφέ του ντόμινο ε, στο Καμερούν ε, δεν, έχει, δεν έχουν εξαφανιστεί οι αντάρτες στη στρατόσφαιρα είναι ακόμα στη γη έχουν κάτι κάνει εκατοντάδες χιλιόμετρα στην στην ε, Ήπειρο για να πάνε να κάνουν τα ίδια κάπου αλλού. Το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει περιφερειακή διάσταση ε, και το λέω αυτό στο πλαίσιο των προσπαθειών σας, τις οποίες θεωρούμε αξιέπαινες για το state building, για την οικοδόμηση κρατικών υποδομών, την ανάπτυξη κρατικών υποδομών. Μην ξεχνούμε ότι έχει το μεγαλύτερο ποσοστό γεννήσεων και το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας κάτω από τα 50. Άρα λοιπόν όλα πρέπει να τα, σχεδόν, να τα κάνουμε σχεδόν από την αρχή σε αυτή την περιφέρεια. Τρίτο στοιχείο. Στη... Στον οδικό σα χάρτη, στο χάρτη πορεία σα, ε, θέλω να επιμείνω σε ένα πράγμα. Όταν μιλάμε για τη διαμεσολάβηση, εντάξει, οι ε, κάτοικοι του Μαλή πρέπει να κάνουν την, πρόταση, την, ε, την επιλογή του. Δεν μπορούμε να μάθουμε τίποτε στους Αφρικανούς, αλλά ελπίζουμε στις διαπραγματεύσεις που θα έχετε μαζί τους να μπορέσετε να τους πείσετε να να μην θεωρούνται όλοι οι Τουαρέγ στο βορρά ε, ε, ε, υπεύθυνοι. Ε, αντιθέτω, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, τους οποίους πρέπει να τους υποστηρίξουμε, δεν πρέπει να τους απομονώνουμε. Και τελευταίο, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό όλων των αναγκών και ότι θα ήταν σημαντικό να κάνουμε μια νέα συνάντηση τη, στο επόμενο διάστημα για να συζητήσουμε τις ανάγκες και για να κάνουμε πράξη ό,τι χρειάζεται σε περιφερειακό επίπεδο. Αν χρειάζεται, χρειάζεστε πολιτική ε, ε, υποστήριξη, ευχαρίστως ε, να σας βοηθήσουμε. Ε, αν ε, δεν έχουμε, αν δεν έχετε άλλους ε, συμμάχους, είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε να σας βοηθήσουμε και θα ήταν χαζό να μην σας υποστηρίξουμε. Η υποστήριξή μας δεν θα είναι μία μεμονωμένη δράση, αλλά θα μπορεί να αποτελέσει τμήμα της γενικότερης βούλησης να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και κλείνει το μικρόφωνο. Sans Χωρίς να καθυστερούμε θα περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης ε, που είναι το εξή. Στην τελευταία μας συνεδρία είχαμε ανταλλαγή απόψεων για τα, των πιλωτικών προγραμμάτων ε, στον ανθρωπιστικό εθελοντισμό που υπάρχουν από το 2011 ε, η συγκήτρια είναι υποφαινόμενη μετά από πολλές διαβουλεύσεις όπως επίσης και με τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Σήμερα σας παρουσιάζουμε την έκθεση που πρέπει να ε, ψηφίσουμε επί τη βάση των διαπραγματεύσεων του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο τριμερούς διαλόγου ανεπίσημου με το Συμβούλιο. Σας παρουσιάζω λοιπόν τι βασικέ ε, γραμμέ τη εκθεσή μου. Δίνω λοιπόν το λόγο στον εαυτό μου, τι πρακτικό. Αγαπητοί συνάδελφοι, Είχαμε ήδη δύο συζητήσει σε σχέση με την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ίδρυση ενό εθελοντικού ανθρωπιστικού σώματο Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πω αυτά που ήδη είπα σε αυτές τις, ε, σε αυτές τις, ε, ε, Συμφωνώ με τους στόχους και τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρότασή της. Όμως κάποιες από τις διατάξεις προτάσεις είναι λίγο αόριστες και πρέπει να συμπληρωθούν και να διευκρινιστούν. Γι' αυτό προτείνω πολλές τροπολογίες για να εξασφαλίσουμε την πραγματική προστιθέμενη αξία της πρότασης ο προβληματισμός, ε, οι σκέψεις ε, γύρω από τις γενικές, ε, για τις γενικές γραμμές της εκθεσής μας βασίστηκαν στην ιδέα του πιλωτικού προγράμματος. Προτείνουμε να αποκλείσουμε τις ένοπλες σειράξεις και, τον, και τα εσωτερικά προγράμματα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των εθελοντών. Στο πλαίσιο των θεομηνιών πρέπει να συμμετέχουν μόνο προς, ως προς την ενίσχυση της ε, ικανότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την προετοιμασία των φυσικών καταστροφών, την πρόληψη αυτών, ε, τη διαχείριση του κινδύνου και τη σχέση μεταξύ του, των, ε, της ε, επίγουσας κατάστασης, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης. Πρέπει να υπάρχει μια πραγματική προστιθέμενη αξία και πρέπει να βασίζεται η ανάπτυξη των εθελοντών στις ανάγκες που αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν επιτόπου ή ήδη ε, υπάρχει αυτός ο στόχος ε, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να είναι ένα καθαρά ανθρωπιστικό ε, σώμα με όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση των ε, προβλεπόμενων ε, οικονομικών πόρων. Πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση της ε, αξίας της ανθρωπιστικής αυτής προσπάθειας και να λάβει υπόψη τη σχέση κόστους-οφέλους. Οι δείκτες που προτείνονται για την αξιολόγηση αυτή είναι μόνο ποσοτικοί, κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό τουλάχιστον ένας ποιοτικός δείκτης πρέπει να υπάρχει για κάθε στόχο επιχειρησιακό, ώστε ο στόχος αυτός ε, να μπορεί να υπάρχει ως τμήμα του νομοθετικού κειμένου. Η ανθρωπιστική συνεισφορά ε, των εθελοντών και η ποιότητα των δράσεων πρέπει να αξιολογείται. Επίσης προτείνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί ένα απλό σύστημα ε, ένα σύστημα πιστοποίησης για τους οργανισμούς αποστολής, συνεργασία όχι μόνο με εταίρους αλλά και ε, με τα ανθρωπιστικά πρότυπα που ήδη υπάρχουν για να μην υπάρχει μεγάλος διοικητικός, ε, διοικητικό άχθος για, τις, ε, για τους μικρομεσαίους οργανισμούς. Πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη τεχνογνωσία και συγκεκριμένη εμπειρία. Πρέπει η επιλογή να γίνεται βάσει συγκεκριμένων προσόντων και βάσει ανταπόκριση σε συγκεκριμένους στόχους. Προτείνω οι εθελοντές ε, να θεωρούνται πιστοποιημένοι ε, εθελοντές ε, της βοήθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναφέρονται σε ένα μητρό το οποίο θα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποστηρίζει όλες αυτές τις, πράξεις, τις δράσεις αξιολόγησης, αναγνώρισης για να, μπορέσουν να δουν, για να μπορέσει να δει τι επαγγελματικά προσόντα χρειάζονται Ε, όσοι ήδη συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας δεν θα έπρεπε να αποτελέσουν τμήμα και αυτού του εθελοντικού σώματος. Ε, πιστεύω ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το οποίο σκοπό έχει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Και τέλος, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σεβάστηκε πλήρως το, τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκ της ε, συνθήκης ε, της ε, Λισαβόνας σε σχέση με τις κατεξιοδότης συμπράξεις. Εμείς προτείνουμε η Προτάσει Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ληφθούν υπόψη σε αυτό το πλαίσιο των νέων προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πολιετές, οι ε, πολιετής στόχοι ε, θα είναι αντικείμενο πράξεων ε, κατεξιοδότηση και όσον αφορά τους στόχους και όσον αφορά τη μεθοδολογία, τους τρόπους εφαρμογής, όπως επίσης και το συνολικό κόστος. Ο προγραμματισμός θα ε, αποφασίζεται με τη διαδικασία των επιτροπών ε, και θα, ε, αναφέρουν την περιγραφή της δράσης όπως επίσης και το αντίστοιχο κόστος αυτής. Ευχαρίστως να ακούσω τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 26 Φεβρουαρίου, 5 η ώρα το απόγευμα. Κύριε Κόρτες Λάστρα. Ναι, Σα ευχαριστώ. Θα σα μιλήσω εκ μέρου τη κυρία Κρετού που για πρόσωπου λόγου δεν μπόρεσε σήμερα να παραστεί. Και μα λέει ότι έχουμε ένα σωρό βίες συγκρούσει και θεομηνίε που έχουν οδηγήσει σε, σε, σε τραγωδία αυξανόμενη παντού. Οπότε οι εθελοντέ μπορούν να βοηθήσουν όσον αφορά την ανταπόκριση τη Ένωση και συμφωνούμε ότι δηλαδή η εγγύηση που παρέχεται για την ασφάλεια αυτών των εθελοντών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κατά τη γνώμη τη και κατά τη γνώμη νομίζουμε ότι το πιο σημαντικό για την επιλογή αυτών είναι το πώ θα γνωρίζουν ε, την επιτόπου πραγματικότητα και κυρίω τι ε, ανάγκε και τι τοπικέ συνήθειε. Και νομίζω ότι η κατάρτισή του θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με εξειδικευμένου οργανισμού με εμπειρία επί και έτσι μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ε, την, ε, την συμβολή τους και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την ανταλλαγή των καλών πρακτικών ε, όσον αφορά την, την επιτόπου εργασία τους οπότε θα πρέπει να ενισχυθεί ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ευχαριστήσω την κυρία η εισηγήτρια για τόσα έκανε για το έργο που σχετικά με αυτή την έκθεση ευχαριστώ πρόεδρος ευχαριστούμε πάρα πολύ και συμφωνώ 100% με αυτό το οποίο είπατε και προβλέπετε επομένω να προβούμε σε αυτή την αξιολόγηση. Κύριε Νιούτον Ντάν, θέλετε το λόγο. Briefly, Madam President and Madam Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κυρία εισηγήτρια υπό τις δύο σας ιδιότητες και δεν ξέρω αν μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτό το πρόγραμμα χωρίς να χρησιμοποιήσουμε ε, την εμπειρία του πιλωτικού προγράμματος. Δεν ξέρω τι πρεσβεύεται, ε, τέλος να συνεχίσουμε. Αλλά έχω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι εν ώψη αυτής της συνάντησης της κορυφής ε, του ΕΜ για το πολιετές πλαίσιο, το χρηματοδοτικό, συνάντηση κορυφή με όλου του ηγέτε. τι, γίνεται με το, το, αποκύημα αυτή τη συνάντηση, πώ θα επηρεάσει αυτό που συζητάμε τώρα, γιατί θα πρέπει να δούμε το ότι το Συμβούλιο θέλει να περικόψει την πρικοδότηση αυτού του προγράμματος. Μήπως θα πρέπει να δώσουμε μάχη. Ναι, ναι, σίγουρα. Και για τον αγώνα αυτόν υπολογίζω και στη βοήθειά σας για αυτές τις περικοπές της δημοσιονομικής. Πάντως προς το παρόν δεν ξέρουμε τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρω μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας βοηθήσει για ενημέρωση. Κυρία, κύριε, ο κύριο Γιάνν Κλάρκ. Um, um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επί του προκειμένου, δυστυχώς δεν μπορώ να σας ενημερώσω σε αυτή τη φάση. Έτερον, έτερος, καλά. Ούτε θέλει κανεί το λόγο. Α, η Επιτροπή θέλει κάτι να πει. Um, first, uh, thank you very... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε για την έκθεση. Ε, πάρα πολύ θετικό. Ε, είναι κάτι το οποίο βοηθά την πρωτοβουλία μας και πολλές από τις ε, τροπολογίες και πάρα πολύ σημαντικές γιατί ξεκαθαρίζουν, βελτιώνουν, φωτίζουν το κείμενο. Και έχω κάποια θέματα είναι κάποιο σημείο μας προβληματίζουν, πρέπει να σας αναφέρω και κυρίως ε, σε σχέση με όσα είπατε εσείς για τον πολιετή προγραμματισμό αυτής της πρωτοβουλίας, κάτι το οποίο σχετίζεται με την τροπολογία 46. Οπότε και εμείς κάπως προβληματιζόμαστε σε αυτό το σημείο, γιατί ε, εδώ δεν πρόκειται περί του μέσου αναπτυξιακής εργασίας ε, ή ε, του, του, μέσου, της ε, γειτονίας, τέλο πάντων δεν είναι, δεν είναι θέμα τέτοιο χρηματοοικονομικό. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα γίνει θεομηνία, πότε θα έχουμε ανθρωπιστική ε, κρίση. Μέσω πρόθεσμα δεν υπάρχουν τέτοια προγνωστικά. επομενω αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να συνειδητοποιήσουμε πόσο αλλάζουν μέρα τη μέρα οι, οι σε αυτό το μέτωπο. Γι' αυτό και λέμε αυτά σχετικά με τον πολιτικό προγραμματισμό. Δεν νομίζω ότι ο στόχος, η φύση του προγράμματος εξυπηρετείται κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί πρόκειται για μικρό χρηματοδοτικό μέσο σε σχέση με κάποια άλλα τα οποία αφορούν εξωτερική δράση. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι αυτό θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, οπότε και ε, προτιμούμε η πρόταση να μείνει όσο έχει με τα αιτήσια αυτά προγράμματα. Και έχουμε άλλωστε αυτό το επταετές μέσω πρόθεσμο προγραμματισμό. Και τώρα, κάτι άλλο το οποίο μπορεί να ανακύψει αφορά αυτά τα καταπιστεύματα. Όπως ορίζει η τροπολογία 47. και όλα αυτά περνάνε μέσα από ζυμώσεις τριμερεί των τριών των οργάνων, οπότε και το πιο σωστό είναι να δούμε τι θα προκύψει από αυτόν τον, τον τριμερή διάλογο, την τριμερή συνάντηση. Και να δούμε αυτή η πρωτοβουλία τι επιπτώσεις θα έχει. Επίσης, δεν είναι σωστό το ότι θέλουμε τις νέε χώρες να τις εξαιρέσουμε από αυτή την πρωτοβουλία έχουμε ήδη προτείνει να υπάρξει κάλυψη των υποψηφίων χωρών σε σχέση με τη γενικότερη πολιτική της, της Κομισιόν για να ξανοιχτούμε προς αυτές τις χώρες και τα πολιτιστικά κλπ. Και, και γενικά, πρόκειται έχει κάποια γενικευμένη πρακτική. Επομένως, ε, και στο πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίε να δούμε κατά πόσον αυτές οι χώρες θέλουν να συμμετάσχουν, τότε να δούμε πώς δεν θα υποστούν τις συνέπειες των περικοπών του προπολογισμού και να δούμε κατά πόσον θα υπάρχουν κάποια κονδύλια τα οποία να διτεθούν για αυτές τις χώρες. Ή αν δεν θα χρησιμοποιηθεί ο κάθε αυτό προπολογισμό. Κάτι άλλο τώρα το οποίο θέλω να σας δείξω συντομία για, για την τροπολογία 52 όσον αφορά τον παρατηρητή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτές τις ε, διαδικασίες Επιτροπής οι οποίες ήδη ε, διέπονται από έναν κανονισμό του 2011 και το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα του ελέγχου και προσβασιμότητα σε όλα τα έγγραφα, αλλά όχι αναγκαστικά ως παρατηρητής. Και επομένως αφού έχουμε αυτόν τον κανονισμό δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Επίσης, συμφωνούμε με εκείνες τις τροπολογίες οι οποίες σχετίζονται με την μη ανάπτυξη εθελοντών εκεί που υπάρχει ενόπλη σύγκρουση. Επίσης αναφέρεται στην τροπολογία ε, το θέμα των εσωτερικών συγκρούσεων αν, ε, αναταραχών. Ε, έχουμε έρθει σε επαφή με τους νομικούς μας συμβούλους οι οποίοι είπαν ότι αυτό το internal disturbances είναι όρος αγγλικός στο αγγλικό κείμενο. Δεν υπάρχει σε άλλες μεταφράσεις του κειμένου. Ε, δεν είναι όρος δόκιμος του, είναι εξονομικός όρος, δεν, είναι θέμα, δεν είναι όρος του διεθνούς δικαίου. Οπότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσο εδώ καλύπτονται οι ένοπλες συγκρούσεις ή οι μη διεθνείς ε, ένοπλες συγκρούσεις. Οπότε να δούμε κατά πόσο θα καλύπτονται και ο εμφύλιος. Επίση έχουμε την τροπολογία έχουμε 16, εκεί που προτείνεται συγκρότηση κάποιου βήματος, κάποιου φόρουμ διαβούλευσης. Μήπως αυτό θα έπρεπε να θυγεί στα πλαίσια αυτού του δικτύου που προτείνει ο κανονισμός, τόσο ώστε να μην έχουμε επιπλέον πολλά ε, φόρα. Οπότε ίσως να εξετάσουμε το ρόλο του δικτύου θα μπορούσε να επεκταθεί για να καλύψει και τα της διαβούλευσης, αυτά τα οποία προτείνει αυτή η διαβούλευση. Και να μην συγκροτήσουμε ακόμα ένα φόρουμ. Επίσης, χαιρετίζουμε αυτούς τους ποιοτικού δείκτες με την ε, προειδοποίηση ότι θέλουμε να μειώσουμε τους δείκτες, να μην έχουν παραπολούς και από πλευρά δημοσιονομική θέλουμε να περιοριστούμε σε τρεις δείκτες αναστόχων. Άρα αν υπάρξουν δείκτες να μείνουμε στο όριο των τριών. Αυτά καταρχήν, αλλά όπως είπα στην αρχή, γενικά θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετική έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα λάβω υπόψη αυτά που είπατε. Ήταν πολλά αυτά τα σημεία. Όντω πρέπει να περιμένουμε τον τριμερή διάλογο. Υπάρχει κάτι επί του οποίου επιμένω. Δηλαδή θέλω να μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ε, πάντως τις παρατηρήσεις σας τις σημείωσα και μαζί με τους συναδέλφους και με τους συνεργάτες ε, θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη συμμετοχή σας. Και περνάμε στο τελευταίο σημείο. είναι η παρουσίαση από τον συνάδελφο Φιλίπ Κατσομαρέκ της έκθεσης σχετικά με την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας στον Άγιο Βικέντιο και τις Γραναδίνες το Δεκέμβριο που μας πέρασε μετά την κοινοβουλευτική συνάντηση στο Σουρινάμ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κασμαρέκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ήταν πολύ μικρή η αντιπροσωπεία. Ε, κάθε φορά μετά από μία μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή χωρών και προσπαθούμε να οργανώνουμε δύο τέτοιες αποστολές. Είχε προγραμματιστεί μία να πάει στις Γρεναδίνες και Άγιο Πικέντιο και η άλλη στην Αγία Λουτσία. Επειδή δεν μπορούσαμε όμως να έχουμε αρκετούς βουλευτές ε, που θα συμμετείχαν και θα ψήφιζαν στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ακυρώθηκε η αποστολή στη Σανταλουτσία και πήγαμε μόνο στον Άγιο Βικέντιο. Και μόνο μία μέρα μείναμε εκεί. Με ιδιαίτερα εντατικό πρόγραμμα όμως. Παρότι αυτή η αποστολή λοιπόν διήρκεσε μόνο μία μέρα, συγκεντρώσαμε πολλές πληροφορίες. Θα έχετε ήδη λάβει τη γραπτή μας έκθεση από αυτού. Ε, κάναμε επαφές υψηλού επίπεδου με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης και του κυβερνώντος κόμματος. Συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, συναντηθήκαμε με τον πρωθυπουργό Γκονζάλες που δεν το είχαμε προγραμματίσει από πριν, αλλά ήρθε εκείνο σε μια συνάντησή μας οικειοθελώς, παρότι ήταν Σάββατο. Και μας αφιέρωσε χρόνο είναι ένας ηγέτης που ξέρει τι θέλει να κάνει και έχει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για τη χώρα του. Ήταν λοιπόν ιδιαίτερα χρήσιμη η συνάντηση που κάναμε μαζί του. Μιλήσαμε και με εκπροσώπους των Υπουργείων Γεωργίας, Υγείας και Περιβάλλοντος με ε, εκπροσώπους από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης επίσης. Λοιπόν, τι να σας πω για τον Άγιο Βικέντιο. Είναι μια οικονομία πολύ μικρής κλίμακας, μια ευάλωτη οικονομία διότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικούς παράγοντες, όπως το κλίμα. Σήμερα μιλήσαμε με την Επίτροπο Χέντεγκορ και μας ανέφερε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μία φυσική καταστροφή μπορεί να κοστίζει 2% του ΑΕΠ μιας χώρας. Στην περίπτωση ε, του Άγιου Βικέντιου, ο τυφώνας Τόμας οδήγησε σε απώλεια 20% του ΑΕΠ. Είναι λοιπόν μια χώρα με μια πολύ ευάλωτη οικονομία, όπου μία και μόνη φυσική καταστροφή μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες. Και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα του Αγίου Βικέντιου. Το δεύτερο μείζον ζήτημα είναι το ότι αυτή η οικονομία δεν είναι πολύ ευέλικτη, δεν είναι διαφοροποιημένη οικονομία, βασίζεται κυρίως στη γεωργία και ιδίως στην καλλιέργεια της μπανάνας. Έχει επίσης και τουρισμό και υπάρχουν και εμβάσματα από ε, κατοίκους εξωτερικού που στέλνουν εμβάσματα πίσω στη χώρα τους. Είναι πάντως μια οικονομία που δεν είναι διαφοροποιημένη. Η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει κάποιες ε, προοπτικές ανάπτυξης για να τονώσει την οικονομία του Αγίου Βικέντιου και ένα πρόγραμμα που είχε επιλεγεί ως στρατηγική σημασίας πρόγραμμα δημιουργεί πολλές ανησυχίες διότι προσπαθούν να κατασκευάσουν ένα σχετικά μεγάλο νέο αεροδρόμιο. Επισκεφθήκαμε εμείς ε, το εργοτάξιο και ε, αυτό το αεροδρόμιο θα αυξήσει τη δυνατότητα υποδοχής τουριστών από 100.000 στις 500.000 ετησίως. Ε, είναι μια χώρα που δεν είναι έτοιμη να απορροφήσει τόσο μεγάλο αριθμό τουριστών. Δεν έχει την απαραίτητη υποδομή για να εξυπηρετήσει τόσο μεγάλο όγκο τουριστών. Επομένως είναι ένα έργο αμφισβητήσιμο και δεν είναι και τόσο διαφανής η κατάσταση. Γιατί μας είπαν πώς χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό, αλλά δεν είναι ξεκάθαρη η δομή χρηματοδότησής του. Ακούσαμε κάτι για τη συμμετοχή της Βενεζουέλας και κάποιων ε, χωρών του Περσικού. Συναντήσαμε και έναν ε, μηχανικό από την Κούβα που δουλεύει και αυτός ε, για αυτό το έργο του αεροδρομίου. Πάντως δεν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και δημιουργούνται πολλές ανησυχίες. Και η αντιπολίτευση έχει αμφιβολίες, αλλά βέβαια το ότι η αντιπολίτευση μιλά ανοιχτά για αυτό το θέμα και για τις αμφιβολίες της, μας δίνει την εντύπωση ότι μιλάμε για μια δημοκρατική χώρα. Δεν υπήρχε πίεση δηλαδή προς ε, την αντιπολίτευση να συμφωνήσει με την άποψη της κυβέρνησης. Ούτε φάνηκε να απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων που είναι αρνητικά για την κυβέρνηση. Ένα άλλο θέμα που ίσως ενδιαφέρει την Επιτροπή μας είναι η παραγωγή μπανάνας. Επισκεφθήκαμε δύο φυτίες μπανάνας, όπου παράγονται μπανάνες με βάση το θεμητό εμπόριο και είναι και αυτός ένας τομέας που μπορεί να αυξήσει την οικονομική αποτελεσματικότητα της χώρας αυτής. Στη Γεωργία πάντως πιστεύω ότι αυτό που χρειάζονται είναι η διαφοροποίηση, γιατί αν αυτή η χώρα αρχίσει να δέχεται περισσότερους τουρίστες θα πρέπει να μην εξαρτώνται τόσο πολύ από τις εισαγωγές, γιατί στον Άγιο Βικέντιο εισάγουν λαχανικά από άλλες χώρες. αλλά καλό θα ήταν να διαφοροποιήσουν την εγχώρια οικονομία, να μην είναι μόνο μπανάνες αλλά και άλλα προϊόντα. Ταξιδέψαμε μέσα στη χώρα σε χωματόδρομους ε, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά της μπανάνας και είναι δύσκολη δρόμοι. Δεν είναι σαν τους δρόμους ε, που βρίσκεται κανείς στην Αφρική. Είναι χωματόδρομοι με πέτρες και χρειάζονται ισχυρά οχήματα που να αντέχουν τέτοιους δρόμους. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της συγχρηματοδότησης της κατασκευής ε, οδικού δικτύου για να μπορούν να είναι περισσότερο προσβάσιμα κάποια τμήματα του νησιού. γιατί η καλλιέργεια μπανάνας γίνεται στις παιδιάδες που δεν έχουν τόσο εύκολη πρόσβαση. Πιστεύω ότι ένα βασικό πρόβλημα που χρειάζεται συζήτηση είναι αυτό που σας ανέφερα, το τεράστιο αυτό έργο του αεροδρομίου. Όσον αφορά άλλα αναπτυξιακά έργα, έχουν κάνει μια διάγνωση οι αρχές για την κατάσταση της χώρας και για πιθανές λύσεις και προσπαθούν να βρουν λύσεις με τη βοήθεια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλη αξία αποδίδουν στη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι όπως μας είπαν οι ίδιοι, δεν ε, νιώθουν να υπάρχει πολιτική πίεση στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ νιώθουν πολιτική πίεση όταν συνεργάζονται με άλλους εταίρους, όπως με τη Βενεζουέλα, παραδείγματος χάρη. Δεν μας το είπαν τόσο ξεκάθαρα, αλλά αυτή ήταν η εντύπωσή μας, ότι αυτό υπονοούσαν. υπάρχει κάποια πολιτική εξάρτηση, ενώ κάτι τέτοιο δεν υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επομένως πολύ θετική όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που βοήθησαν για την οργάνωση της αποστολής μας αυτής, τη Γραμματεία, τις αρχές ε, του Αγίου Βικεντίου και Γραναδίνων, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τους πρέσβεις, τον κύριο Μάικλ Μπάρκοτ, που είναι επικεφαλής στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Μπαρμπάντος, ο οποίος μας συνόδευε συνεχώς. Και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του τα διάφορα θέματα και τις πληροφορίες που λαμβάναμε και μας βοήθησαν πάρα πολύ γιατί είδαμε ότι υπάρχει και διαθεσμική συνεργασία που λειτουργεί σωστά. Μερικέ φορέ έχουμε κάποιε ανησυχίε για το πώ λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση ήταν εξαιρετική η συνεργασία μα και ήταν πολύτιμη η βοήθειά του. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ όλου εκείνου που βοήθησαν στην οργάνωση αυτή τη αποστολή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νάιζερ, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ήταν επιτυχής ε, η αποστολή γιατί ήταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη από τη γραμματεία και η έκθεση του Φίλιπ είναι πραγματικά πολύ ακριβής, οπότε δεν έχω τίποτα να προσθέσω. E e η ΕΕΔ, e όχι, έφυγαν. Καλά. Θα είμαι σύντομη γιατί οι διερμηνείς θα πρέπει σιγά σιγά να αποχωρήσουν. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Καλά, κύριε Κατσμάρεκ, σας δίνω πάλι το λόγο για να συνοψίσετε. Μία ακόμη φορά. Νομίζω ότι λάβαμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στο πλαίσιο της αποστολής αυτής. Ήταν μικρή, αλλά αποτελεσματική. Eh bien, parfait. Donc, euh, Λαμπρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κατσμάρεκ για την παρουσίαση αυτή. Υπάρχει τίποτα στα διάφορα? Όχι. Πολύ καλά. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες στις 18 Μαρτίου από τις 3 6.30 και στις 19 Μαρτίου από τις 9.30 από τις 9 μέχρι τις 12.30 και από τις 3 μέχρι τις 6.30. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Ευχαριστή και τους διερμηνείς. Ε, ευχαριστούμε ε, πολύ και κυρίζω το πέρα συνεδρίας.